Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Καθίστε παρακαλώ γιατί σε ένα λεπτό θα αρχίσουμε. Ladies Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Αρχίζει η Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Ομάδα για το συντονισμό της ε, πολιτικής, ε, της οικονομικής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στα γερμανικά τώρα. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ως Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σώμα που εκπροσωπεί πολίτες στον κόσμο. Έχω την ιδιαίτερη χαρά σήμερα να σας καλωσορίσω όλους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η πρώτη τέτοιου είδους κοινή ε, συνεδρίαση εθνικών και ευρωπαϊκού κοινοβούλιο με βουλευτές λοιπόν από τις Εθνικές Βουλές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προηγήθηκαν συνεδριάσεις τόσο των πολιτικών ομάδων όσο και συναντήσεις με τις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές τις τελευταίες ημέρες. Αλλά ε, ε, ταυτόχρονα θα υπάρξει και συνεδρίαση της Ολομέλειας. Συνεδρίαση λοιπόν των ομάδων, συνεργασία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και ολομέλεια. Χαιρόμαστε όλους ιδιαιτέρως που έχουμε την ευκαιρία να υποδεχόμαστε ε, συνολικά 103 βουλευτές από 26 εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την πρώτη ε, Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα. Μας τιμά ιδιαίτερα η παρουσία τεσσάρων προέδρων Εθνικών Κοινοβουλίων. Ο κύριος Σομπαρέ από την Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ανδρέ Φλαό, πρόεδρος της Βελικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο κύριος Μισελ πρόεδρος της Βουλής της Μάλτας. Ο κύριος Βαλέριος Στέφαν Σκονέα, πρόεδρος ε, της Ρουμανικής Βουλής. Καλώς ορίσατε θερμά. Επιπλέον, έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίζουμε 30 προέδρους ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών, όσο και 16 αντιπροέδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών. Χαιρόμαστε λοιπόν για την παρουσία όλων των βουλευτών των Εθνικών Κοινοβουλίων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μαζί με εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και επισήμους. Ε, καλωσορίζουμε σήμερα ε, και το λέω δημόσια 185 ε, συμμετέχοντες από εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι αριθμός εντυπωσιακός και υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των θεμάτων που θέλουμε να συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα, αλλά και του τρόπου που αποφασίσαμε της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας και μακάρι να είναι ευκαιρία αυτή για να δώσουμε μια κοινή απάντηση στην πρόκληση και στην απέτηση του άρθρου 13 της συνθήκης για τη συνεργασία Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την σύσφυξη ε, των σχέσεων Ελπίζω αυτό το πρότυπο της ε, εβδομάδας ε, που επιλέξαμε να ε, πριτανεύσει και να δοθεί και συνέχεια με τους Προέδρους των Κοινοβουλίων τον Απρίλιο στην Κύπρο. Ποια είναι τα βασικά μας μελήματα και η ουσιαστική ανησυχία της συνάντησης αυτής. να τονώσουμε τη δημοκρατική πτυχή και διάσταση του ευρωπαϊκού εξαμήνου και της οικονομικής πολιτικής. Προσπαθούμε και εδώ ε, στο Κοινοβούλιο επίσης να ε, τονίσουμε και ε, το συντονισμό της κοινωνικής πολιτικής. Πρωταρχικός στόχος του ευρωπαϊκού εξαμήνου ποιος είναι. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα πρέπει εκ των προτέρων να δέχονται έναν προσανατολισμό σε θέματα οικονομίας. Και γενικά στόχος είναι ο συντονισμός των οικονομικών και των κοινωνικών πολιτικών όσο και των δημοσιονομικών πολιτικών ε, στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτικής όπως είναι η φορολογική πολιτική και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Να βελτιωθεί λοιπόν αυτή η συνεργασία. Από κοινού θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιρροή μας και τις δυνατότητες που έχουμε. Τα Εθνικά Κοινοβούλια απέναντι στις κυβερνήσεις τους σε ευρωπαϊκά θέματα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλους τους τομείς όπου η Ευρώπη αποφασίζει ως σύνολο, ως κοινότητα. Και όπου υπάρχουν φαιές ζώνες με συναρμοδιότητες, συχνά είμαστε κατακαιρματισμένοι, χρειάζεται ενισχυμένη συνεργασία και συντονισμός. Όλα τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν τους στόχους στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ήδη από τώρα έχουν εκπονήσει εθνικά προγράμματα και στρατηγικές για την οικονομική ανάπτυξη, για την ανταγωνιστικότητα, για την κοινωνική συνοχή, αλλά και ε, για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Για να ενισχυθούν σε αυτές οι προσπάθειες όμως δεν αρκούν οι προσπάθειες μεμονωμένων κρατών μελών. Για να φτάσουμε στους στόχους αυτούς χρειάζεται ακριβώς στοχευμένη συνεργασία και συντονισμός αυτών των προσπαθειών. Αυτό είναι κομβική σημασία για να επιτύχει και χρειάζεται ενίσχυση των κοινοβουλίων ε, κατά τη διάρκεια της λήψης των αποφάσεων και της διαμόρφωσης αυτών των αποφάσεων. Και υποθέτω ότι και για σας όπως και για μένα έχει σημασία και υπάρχει και σύνδεση μεταξύ ε, της ετήσιας έκθεσης ανάπτυξης, ε, των, κοινωνικέ ε, κοινωνικές πολιτικές, κατευθυντήριες γραμμές, το six το λεγόμενο τη δέσμη των έξι οδηγιών, το two που ακολούθησε και το σύμφωνο για τη σταθερότητα την Οικονομική Ένωση και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και τον προϋπολογισμό. Όλα αυτά είναι για μένα άρρηκτα συνδεδεμένα. Μέχρι τις 15 Απριλίου θα πρέπει να έχετε διαβιβάσει οι κυβερνήσει τα εθνικά του σχέδια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλη Μαΐου θα δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστάσεις ειδικέ ανά χώρα. Και ε, ξεχωριστές συστάσεις για την Ευρωζώνη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έρθει να τα εγκρίνει όλα αυτά τον Ιούνιο και το επόμενο βήμα ε, είναι το Συμβούλιο Υπουργών τον Ιούλιο βάσει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθεί να τα εγκρίνει όλα αυτά και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα σχέδια προϋπολογισμού. Έτσι λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. όλες αυτές οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες, οι στόχοι, πώς συνδέονται με όλα αυτά τα μέτρα. Από την ετήσια έκθεση, την οικονομική, την αναπτυξιακή, μέχρι τις κοινωνικές ε, κατευθυντήριες γραμμές, το ΣΥΚΣΠΑΚ, το ΤΟΥΠΑΚ και την ίδια τη συνθήκη και το Σύμφωνο Σταθεροποίησης, η σταθερότητα συντονισμού και ε, της ΟΝΕ και του προπολογισμού και των δημοσιονομικών πρόπτικων. Πώς συνδέονται όλα αυτά, πώς κουμπώνουν μεταξύ τους. Αυτό χρειάζεται ένα στενό συντονισμό. Και βεβαίως και σωστά έτσι εδώ ενισχύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλέσαμε λοιπόν ένα τμήματάρχη και ε, ομιλητές και ε, ε, καλωσορίζω τον κύριο Ευρώ στο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Όλι Ρεν, που είναι αρμόδιος για οικονομικά και νομισματικά θέματα για την ΟΝΕ. Επίσης καλέσαμε τον αρμόδιο επίτροπο για θέματα κοινωνικά, απασχόλησης και ε, κοινωνική συμπερίληψη που είναι ο κύριος Λάσλο Άντο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ να συζητήσουμε ε, και να εμπλουτίσει τις εργασίες μας με την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με τη μορφή της ίσιας έκθεσης ανάπτυξης ε, καλείται αυτή η έκθεση να βοηθήσει ε, τη συνεργασία και τη στρατηγική μας στα κράτη-μέλη αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2013. Προσθέτω αμέσω ότι μια τέτοια κοινοβουλευτική ε, εβδομάδα δεν θα πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο ε, επαφορμή ε, την ετήσια αυτή έκθεση, αλλά και το φθινόπωρο χρειαζόμαστε μια αντίστοιχη για τον προπολογισμό. Στο τέλος του συζητήσεως σήμερα το πρωί θα συνεδριάσουν οι επιτροπές οικονομικών, ανάπτυξης, απασχόλησης μάλλον και προϋπολογισμού για να ασχοληθούν με τα επιμέρους ζητήματα και τις λεπτομέρειες που ε, τις αφορούν. Εδώ στο Προεδρείο έχουμε και τους Προέδρους των Αρμόδιο Επιτροπό. Ο κύριος Λαμασούρη είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ε, η κυρία Μπόλς είναι Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και η κυρία Περμάς Μπερές είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε ε, για τη συμμετοχή σας και τις συζητήσεις. Ποιος είναι ο στόχος, λοιπόν, να συζητήσουν τα συμπεράσματα οι επιτροπές και την Τετάρτη το πρωί να υποβληθούν όλα αυτά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Ε, συζήτηση για το θέμα αυτό έρχεται σε μια στιγμή επίκαιρη. Δεν θέλουμε να αρρωποιήσουμε, αλλά ούτε να δραματοποιήσουμε την κατάσταση. Ε, είναι παραμονές της ε, Συνόδου Κορυφής, του Συμβουλίου και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και ως συγκυρία. Με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχουμε νέες αρμοδιότητες για τη χάραξη ε, της πολιτικής και της προτεραιότητας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και εμείς οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την αλλαγή και να τους δώσουμε την απαραίτητη δημοκρατική νομιμότητα με τη δική μας διαμόρφωση των εξελίξεων. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει και στο μέλλον να ενισχυθεί. Για πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν προτάσεις δόν σε όλους τους τομείς πολιτικής που μας αφορούν. Ιδιαίτερα στις χώρες που ακολουθούν προγράμματα ε, υπάρχουν συστάσεις λεπτομερείς αναχώρα που δίνουν το πλαίσιο για τις απαραίτητες ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μέτρα οικονομικής πολιτικής. Και όλα αυτά είναι προαπαιτούμενες δράσεις ε, για ε, να φτάσουμε στους στόχους μας της Ευρώπης 2020. Ταυτόχρονα επαναλαμβάνεται μια συζήτηση περί δημοκρατικού ελλείμματος ως προς το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Ε, τουλάχιστον ως προς τη λήψη των αποφάσεων και τη διαδικασία τους. Περί τίνος πρόκειται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο διακυβερνητικό και κλεισμένο των θυρών μετά από προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα, είναι δύσκολο μεταξύ άλλων να εντοπίσουμε ποιος αποφασίζει τους στόχους αυτούς πολιτικής και ποιος τελικά φέρει και την ευθύνη για αυτούς. Σε τελική ανάλυση, εμείς έχουμε την ευθύνη για την εφαρμογή ε, των ε, αποφάσεων που λαμβάνονται από κοινού. Γι' αυτό λοιπόν σε εμά αναπόκειται τους εκλεγμένους εκπροσώπους των λαών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στα Εθνικά Κοινοβούλια όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να φροντίσουμε να βρούμε τους κατάλληλους δρόμους για να συνοδεύουμε και να πλαισιώνουμε τις αποφάσεις, ε, τις οικονομικές και τις δημοσιονομικές που δεν σταματούν πλέον στα εθνικά σύνορα. Έχουμε μια πρόκληση στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε και αυτή η πρόκληση είναι ευρωπαϊκή. Ο καθένας από εμά φέρει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική διάσταση που να παρακολουθεί αυτές τις διαδικασίες και τις εξέλιξεις. Και εδώ υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει ακόμα να αντιμετωπίσουμε και πολλά ερωτήματα να απαντήσουμε. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει με ακρίβεια να διαμορφώσουμε τον τρόπο συνεργασίας εθνικών ε, με Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ορίζει το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο ε, για τη συνεργασία αυτή. Βεβαίως έχετε συζήτηση αυτό, αλλά θα σας παρακαλούσα να καταλάβουμε ότι η σημερινή και αυριανή μας συνεδρίαση δεν έχει αυτό το αντικείμενο. Και δεν θα πρέπει να μας ε, κάνει να λησμονούμε ότι υπάρχουν και θέματα δημοσιονομικά πίσω από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και ακριβώς επειδή ε, το θέμα είναι πάρα πολύ βαθύ, ε, το επόμενο διήμερο θα έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση αυτών των θεμάτων. Πολύ σύντομα τώρα κάποιες παρατηρήσεις κυρίες και κύριοι για τη σημερινή συζήτηση και τα διαδικαστικά. Στην αίθουσα αυτή έχουμε 22 γλώσσες. Μπορείτε να παρακολουθείτε, θέλετε και να ακούτε και να μιλάτε τη μετρική σας γλώσσα. Θα φροντίσουμε να πάρουν το λόγο όσο γίνεται περισσότεροι βουλευτές για να μας παρουσιάσουν τις απόψεις τους. Επειδή όμως έχουμε χρόνο περιορισμένο και μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, σας παρακαλώ ήδη από τώρα να δείξετε κατανόηση. Δεν θα μπορέσει να πάρει το λόγο κάθε βουλευτή σε κάθε συνεδρίαση. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να συμφωνήσουμε ένα περιορισμένο χρόνο αγόρευσης, το πολύ τρία λεπτά αναμιλητή, κατά διάρκεια συζήτηση αυτό το τρίλεπτο μπορεί και να μειωθεί. Στα έδρανά σας ε, έχετε τα λεγόμενα speaking notes cards. Αν θέλετε δηλαδή να ζητήσετε το λόγο σας παρακαλώ να συμπληρώσετε αυτά τα έντυπα και να τα διαβιβάσετε. Στο Προεδρείο έχουμε στην αίθουσα συνεργάτες που θα τα ε, μαζεύουν. Αυτό ισχύει και για τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και για τους ευρωβουλευτές. Εδώ είναι όλοι οι βουλευτές ίσοι. Ε, όποιος θέλει να μιλήσει θα πρέπει να συμπληρώνει αυτή την κάρτα. Και όταν δίνω το λόγο θα τηρώ τον εξή κανόνα. Δύο εθνικοί βουλευτέ ε, και μετά ένα ευρωβουλευτή. Δύο προ ένα δηλαδή. Ένα αλλάξει με αυτή τη σειρά. Είναι λοιπόν σαφή και τα διαδικαστικά. Ωραία. Θα δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Όλη Ρέν. Παρακαλώ, Όλη, έχεις το λόγο. Thank you. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, Ότμαρ. αξιότιμη συνάδελφε Κάρασα. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι αποτελεί τεράστια ευχαρίστηση για μένα το να βρίσκομαι εδώ σε αυτή τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Αυτή η σύνοδος ε, συγκεντρώνει εκπροσώπους ε, τόσο των Εθνικών Κοινοβουλίων όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια συζήτηση περί συντονισμού οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμένου. Πρόκειται για ένα σαφές, ε, ορατό βήμα προς την ανάδυση ενός πιο ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου. Το βήμα αυτό εμφανίζεται την κατάλληλη στιγμή. Βρισκόμαστε εν μέσω των προετοιμασιών ε, του φετινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τρίτη φορά που βασίζεται στην ε, στρατηγική Ευρώπη 2020 για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Επίσης ε, βασίζεται στην τελευταία της ανασκόπηση της ανάπτυξης που παρουσίασε η Κομισιόν τον Νοέμβριο. Αναμένουμε ότι αυτές οι προτεραιότητες πολιτικής ε, θα αποτυπώνονται στα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης των κρατών μελών και στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα όπως θα παρουσιαστούν τον Απρίλιο για την ε, αξιολόγηση ομοτήμων του Συμβουλίου και την αξιολόγηση της Κομισιόν. Το βήμα αυτό είναι επίσης ε, έγκαιρο, διότι παρέχει δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία στα κράτη-μέλη. Καθώς βρισκόμαστε στο μέσο της συζήτησης, παρακολουθούμε τη συζήτηση αυτή εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ε, τροποποίησης της θεσμικής, της αρχιτεκτονικής. Τα κοινοβούλια είναι υπόλογα για τις πολιτικές αυτές ε, ενώπιον των πολιτών μας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως τρέφονται οι πολίτες για να βρουν απαντήσεις. Αυτή η τεράστια ευθύνη απαιτεί να βρούμε τον καλύτερο δρόμο προς τα μπρος ε, μέσω μιας ανοιχτής συζήτησης και διαβούλευσης. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας παρουσιάσω σήμερα στην αρχή αυτής της ε, συζήτησης, τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις προτεραιότητες πολιτικής για τη φετινή χρονιά 2013. Πριν από αυτό, ωστόσο, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω που βρισκόμασταν πριν από ένα χρόνο και να κάνω μια σύγκριση με τη σημερινή κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πριν από ένα χρόνο βρισκόμασταν σε βαθιά αβεβαιότητα για την Ελλάδα. Υπήρχαν σοβαρές ανησυχίες για την Ιταλία και την Ισπανία. οι ελλείψεις των ε, διαδικασιών ρευστότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτυπώνονταν στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα και θα θυμάστε ότι ακούσαμε αμέτρητες προφητείες, κασάνδρες που προέβλεπαν ε, τη διάσπαση της Ευρωζώνης. Η περσινή χρονιά όμως, το 2012, κατέληξε να είναι μια αποφασιστική χρονιά κατά την οποία η Ευρωζώνη απέδειξε την πολιτική της αντοχή και έλαβε τολμηρές αποφάσεις που διασφαλίζουν την ενότητα και την βιωσιμότητα του ευρώ. Σήμερα όλες αυτές οι προβλέψεις διάσπασης της Ευρωζώνης ε, έχουν εξελευθεί. εντελώς ουσιαστικά από τη δημόσια συζήτηση. Παρά αυτή την ε, πρόοδο Έχουμε να, αντιμετωπίσουμε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις, ε, υψηλή ανεργία, πολύ αργή ανάπτυξη της οικονομίας και έτσι δεν υπάρχει περιθώριο για χαλαρότητα. Χρειαζόμαστε αποφασιστικότητα και έντονες δράσεις ε, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασία. και πρέπει να εργαστούμε σκληρά ώστε οι λαοί τη Ευρώπη να αντιληφθούν ότι απαιτούνται αυτές οι πολιτικές ώστε να διατηρηθεί δυνατή η οικονομία και η δημοκρατική νομιμότητα αποτελεί το κλειδί για αυτή τη φιλόδοξη πολιτική ατζέντα. Οι προσπάθειές μας ε, εστιάζονται κυρίως ε, στη μεταρρύθμιση και στον εξυγχρονισμό της, ε, του μοντέλου οικονομίας κοινωνικής, οικονομίας αγοράς της Ευρώπης. Υπάρχουν τρεις ροές εργασιών που συνθέτουν ε, την ε, απόκρισή μας στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής. Πρώτον, χρειάζεται να διατηρήσουμε το βηματισμό της οικονομικής μεταρρύθμισης ώστε να υποστηρίξουμε την ε, εξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αυτή η εκ νέου εξισορρόπηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρατηρούμε τη μεταστροφή σε χώρες με ελλείμματα των τροχών των λογαριασμών. Θα σα δώσω μερικά παραδείγματα. Στην Ιρλανδία οι εξαγωγές παρουσιάζουν αύξηση και οι επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ η εγχώρια ζήτηση είναι αρκετά χαμηλή. Ταυτόχρονα όμως η οικονομική ανάπτυξη προχωρά. Παρατηρούμε αύξηση της παραγωγής, βελτίωση της παραγωγής στην Ιρλανδία. Σε άλλες χώρες όπως Πορτογαλία προετοιμάζονται για επιτυχή επιστροφή στη χρηματοδότηση των αγορών όσον αφορά το δημόσιο χρέος τους. Στην Ισπανία η ανεργία είναι πολύ ψηλή, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι εξαγωγές. Ο όγκος των εξαγωγών στην Ισπανία είναι υψηλότερος από ποτέ. Ακόμη και στην Ελλάδα, οι απώλειες ανταγωνιστικότητας της τελευταίας δεκαετίας ε, καλύπτονται σιγά σιγά. Στο μεταξύ και οι χώρες με πλεονόσμα συμβάλλουν σε αυτή τη ε, διαδικασία εξισορρόπησης μέσω του ανοίγματος των αγορών υπηρεσιών, αυξάνοντας την ε, συμμετοχή της, εργασ... της αγοράς εργασίας και βοηθώντας την ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα. Στη Γερμανία παρατηρούμε στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων παρατηρούμε αύξηση των μισθών κατά 0,5% το οποίο θα βοηθήσει την εξισορρόπηση της ε, οικονομίας στην Ευρώπη. Αλλά αυτή η εξισορρόπηση δεν είναι αρκετή. Πρέπει να παραμείνει η ευρωπαϊκή οικονομία παγκόσμια ανταγωνιστική. Δεν μπορεί να επιτρέψει απώλειες ε, στις ε, αγορές στις αγορές ομολόγων όπως είδαμε στην ε, Γαλλία, στη Φιλανδία και στο Βέλγιο. Το δεύτερο σημείο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε ή μάλλον να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, τόσο της μεταπηγητικής βιομηχανίας όσο και των υπηρεσιών. Χθες βρισκόμουν στη Μαδρίτη, στην ε, σύνοδο της τέταρτης επαιτίου της ε, Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων και εκτός από τα δικαιώματα των εργαζομένων, τέθηκε και το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της δυναμικότητας. Αυτά αποτέλεσαν σημαντικά ε, σημεία, σημαντικές ανησυχίες και κατά την άποψή μου πολύ σωστά για αυτό το λόγο πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχητικές απώλειες ανταγωνιστικότητας που παρατηρούνται σε πολλές χώρες οι οποίες ε, μεταφράζονται σε διαρθρωτικές ανεργίες και σε ε, μείωση της, ε, των δυνατοτήτων των αγορών. Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. Την τελευταία δεκαετία μεταξύ 2000 και 2011 συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργασίες ε, απολέστηκαν στον τομέα της μεταπίσης σε διάφορες χώρες και 750.000 θέσεις στον τομέα της μεταπίσης στην Ισπανία. ως αντίδραση σε αυτή την τάση τα υψηλά επίπεδα χρέους, η γρήγορη γύρανση του πληθυσμού και το γεγονός ότι πάνω από τις μισές κοινωνικές δαπάνες σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα ε, είναι ευρωπαϊκές. Ε, βλέπετε τι φορτίο έχει να φέρει η ευρωπαϊκή παραγωγική οικονομία για να υποστηρίξει το κοινωνικό μας μοντέλο. Αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αγαπάμε να ζούμε. Αγαπητοί φίλοι, θα πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την τάση. Η Ευρώπη πρέπει να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητά της. Αυτό δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική διάσταση. Σημαίνει βιώσιμη αυξή της ε, κοινωνικής ε, ε, πολιτικής. Και πιστεύω η οποία θα βοηθηθεί από την ανάπτυξη. Και πιστεύω ότι αν συνεχίσουμε τι μεταρρυθμίσει, όχι για να κάνουμε μεταρρυθμίσει, αλλά μεταρρυθμίσει για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασία, μεταρρύθμιση για ενίσχυση τη ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία. Τι χρειάζεται λοιπόν για να δημιουργήσουμε θέσει εργασία και να ενισχύσουμε την παραγωγικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Χρειαζόμαστε υποστήριξη, έρευνα και καινοτομία, καθώς και εκπαίδευση και κατάρτιση. Χρειάζεται να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και τις ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειάζεται να ολοκληρώσουμε την οικονομική επισκευή εντό εισαγωγικών ώστε να βοηθήσουμε τις πιστώσεις προς ε, νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις δημόσιες επενδύσεις όπως κάναμε πρόσφατα με την ε, ε, κεφαλαϊκή ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πρέπει να δημιουργήσουμε έξυπνες, έξυπνους κανονισμούς που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη Επίσης πρέπει να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις ε, στις ε, αγορές εργασίας μας. Εξισορροπημένες αλλά φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις που θα βοηθήσουν στην άρση των εμποδίων δημιουργίας θέσης εργασίων, που θα διευκολύνουν τη δημιουργία μόνιμων συμβολέων εργασίας, που θα διασφαλίζουν ότι όσοι χάνουν τις δουλειές τους σε περίοδους ύφεση μπορούν να υπολογίζουν σε μια πραγματική υποστήριξη ώστε να επιστρέψουν στις θέσεις, στην αγορά εργασίας ή στην κατάρτιση. Μεταρρυθμίσεις που θα σέβονται ε, τη συλλογική, το συλλογική, τη συλλογική φιλοσοφία των χωρών μας. Και εδώ υπάρχει στενή σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμενο. Για ποιο λόγο, διότι η πρόθεσή μας είναι και ελπίζω να συμφωνήσετε ότι αυτά είναι τα κλειδιά για την Ευρώπη, για την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων στην Ευρώπη, θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Αυτού του είδους οι μεταρρυθμίσεις θα αντικατοπτρίζονται στις ε, συστάσεις αναχώρα που θα δοθούν φέτος και εκεί θα εστιαστεί το ευρωπαϊκό εξάμενο σύμφωνα με τα όσα παρουσιάσαμε στην ετήσια ανασκόπηση της ανάπτυξης. Αποτελεί ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα του πώς το ευρωπαϊκό εξάμεινο μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και εγώ υπολογίζω ιδιαίτερα στη δική σας υποστήριξη για την επίτευξη αυτών των στόχων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το τρίτο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι το δημοσιονομικό. Πρέπει να επιμείνουμε σε διαρκή δημοσιονομική εξυγίανση. Σοβαρές ακαδημαϊκές έρευνες και ε, συμπεράσματα εμπειρίας ε, δείχνουν πώς επηρεάζεται η ανάπτυξη από το δημόσιο χρέος δείχνουν ότι όταν φτάνει το δημόσιο χρέος σε επίπεδα του 90 με 100% επηρεάζει πολύ αρνητικά την οικονομική ανάπτυξη, την παρασύρει προς τα πίσω. Δυστυχώς στην Ευρώπη την τελευταία τετραετία το επίπεδο δημοσίου χρέους μας αυξήθηκε από περίπου 60% σε σχεδόν 90% φέτος και του χρόνου αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη. Δεν υπάρχει άλλη Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε έξυπνη και βιώσιμη εξυγίανση. Δημοσιονομική εξυγίανση. Είναι σημαντικό ωστόσο η δημοσιονομική εξυγίανση να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις χώρες, σύμφωνα με το περιβάλλον των χωρών αυτών και την κατάσταση ανάπτυξης του κάθε κράτους μέλους. Γι' αυτό το λόγο χορηγήσαμε παράταση της διόρθωσης υπερβολικού ελλείμματος ε, για ορισμένες χώρες ήδη πέρυσι, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Πράγματι τα δημοσιοοικονομικά στην Ευρώπη βελτιώνονται σταδιακά. Παρατηρούμε τώρα τα αποτελέσματα της δέσμης 6 ε, μέτρων, του Six Pack και της ενισχυμένης οικονομικής διακυβέρνησης το 2009 και 2010. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα στην Ευρωζώνη ήταν μεταξύ 6 και 7% του ΑΕΠ. Πέρυσι μειώθηκαν σε λίγο πάνω από το 3% του ΑΕΠ και αναμένουμε περαιτέρω μείωση φέτος σε περίπου 2,5% του ΑΕΠ. Τέλος, για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και να ξαναβάλουμε την Ευρώπη σε αναπτυξιακή πορεία, θα πρέπει να πείσουμε τους πολίτες μας, καθώς και τις αγορές, όσον αφορά τις πρόπτικες του ευρώ, τις μακροπρόθεσμες πρόπτικες. Πρέπει να οικοδομήσουμε εκ νέου την οικονομική και νομισματική μας ένωση Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα ε, υπόδειγμα με τις προτάσεις της για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και οι προτάσεις της αντικατοπτρίζονται, θα αντικατοπτριστούν και στο έγγραφο του Χερμάν Βαντρόμπεϊ επί του ίδιου θέματος. Δεν προλαβαίνω αυτή τη στιγμή να μπω σε ε, λεπτομέρειες ε, αυτού του blueprint, αυτού του υποδείγματος, αλλά θα σας έλεγα ότι περιλαμβάνει διαδικασίες για την ολοκλήρωση της οικοδόμησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, βραχυπρόθεσμα, δηλαδή σε διάστημα 6 με 18 μήνες από τώρα θα δούμε συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο των τρέχουσών συνθήκων. Ξεκινώντας με την Τραπεζική Ένωση και ως επόμενο βήμα την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού επίλυσης. Αυτό θα αποτελέσει προτεραιότητα κλειδί για φέτος. Φέτος λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο που αφορά τον ο μηχανισμό επιτήρησης για τις ευρωπαϊκές τρέπεζες και η νομοθετική πρόταση για ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό επίλυσης διαφορών επειδή η επιτήρηση και η επίλυση θα πρέπει να συνάδουν. Ευρωπαϊκή εποπτεία και επίλυση. Όσον αφορά τώρα την υποστήριξη των διαρθρωτικών αλλαγών και της δημοσιονομικής εξυγένσης. Αυτά απαιτούν τεράστιες προσπάθειες. Για αυτούς τους λόγους ακριβώς σε αυτό το έγγραφο προτείνουμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού σύγκλησης και ανταγωνιστικότητας ως εργαλείο αλληλεγγύης εντός της Ευρωζώνης. Στόχο θα έχει να υποστηρίζει αποτελεσματικά τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη και να συνδυάζει μια δέσμευση των κρατών μελών για συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις με οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίησή του. Το μέσο αυτό λοιπόν θα χρησιμεύει ως κίνητρο για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και θα βοηθά στην κάλυψη των βραχυπρόθεσμων κόστων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη ολοκλήρωση με αλλαγέ ενδεχομένω των συνθήκων και εδώ θεωρούμε ότι οι κατευθυντήρε αρχέ θα είναι ω εξή. Σε κάθε βήμα προ περισσότερη αλληλεγγύη και αμοιβαιοποίηση του οικονομικού κινδύνου θα πρέπει να συνδυάζεται με αυξημένη υπευθυνότητα και περαιτέρω μοίρασμα της ε, δημοσιονομικής κυριαρχίας. Θα χρειαστούν ε, τα ανάλογα βήματα προς μια πολιτική ένωση για την ενίσχυση της δημοκρατικής λογοδοσίας. Γνωρίζω ότι είναι πολλές οι απόψεις για αυτά τα ζητήματα στα διάφορα κράτη-μέλη και στα κοινοβούλια. Γι' αυτό το λόγο προσδοκώ σε μια ανοιχτή και δημοκρατική συζήτηση για τη μελλοντική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ολοκληρώσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά όλες τις δυσκολίες ε, έχει πραγματοποιήσει τεράστια άλματα το 2012. Η πολιτική μας ατζέντα για τη φετινή χρονιά το 2013 είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και ουσιαστική. Για να την υλοποιήσουμε χρειαζόμαστε ομαδικό πνεύμα και υπευθυνότητα από όλους μας ώστε να αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη μακροπρόθεσμα και να επιστρέψουμε σε βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι κοινέ μα προσπάθειες θα επικεντρωθούν στη μεταρρύθμιση και στον εξυγχρονισμό του ευρωπαϊκού μοντέλου ε, κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και στην πραγματοποίηση πραγματικής ε, ουσιαστικής πρόοδου σε αυτή την πολιτική ατζέντα για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. η φετινή χρονιά θα αποτελέσει σημαντική δοκιμή για την αξιοπιστία της Ευρώπης σε αυτό το δρόμο προς μια ένωση σταθερότητας, προς περισσότερη αλληλεγγύη και λογοδοσία. Θα πρέπει να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την Ευρώπη στο σωστό δρόμο. Και εγώ θα υποστηρίξω αυτό το στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Αναφερθήκατε στο ευρωπαϊκό μοντέλο της ε, βιώσιμης οικονομίας της αγοράς. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον Επίτροπο Λάσλο Άντορ, Επίτροπο, για, για κοινωνικά θέματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές. Η συζήτηση αυτή στο Κοινοβούλιο έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρώπη. Διότι θα πρέπει να λάβουμε μείζονε αποφάσει στο ερχόμενο διάστημα. Λόγω χάρη για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εύρωστα δημοσιονομικά εργαλεία για να υπηρετήσει τι φιλοδοξίε τη για οικονομική ευημερία και κοινωνική πρόοδο και συνοχή. Θα ήθελα να επικεντρωθώ για τη συζήτηση περί Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στο τι συμβαίνει σήμερα, με λίγα λόγια. Πώς έχει η κατάσταση. Εδώ και κάποιο διάστημα διανύουμε μια κρίση που δεν έχει μόνο δημοσιονομική και οικονομική διάσταση χρηματοπιστωτική, αλλά είναι και μια κρίση εμπιστοσύνης, κρίση αξιών. Για πολλούς το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο φαίνεται ότι τελικά δεν θα δώσει τα κοινωνικά ωφέλη ή την κοινωνική συνοχή που ήλπιζαν. Ταυτόχρονα, αυτό είναι απαραίτητο, απολύτως απαραίτητο. Με την τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκε πριν από δύο εβδομάδες βλέπετε ότι υπάρχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και πολλοί βρισκόνται στο κατόφλι της στόχης του κοινωνικού αποκλεισμού αυτή τη στιγμή. Είναι το 1 τέταρτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Επίσης υπάρχει πόλωση. Πόλωση μεταξύ χωρών που είναι δημοσιονομικά σταθερές και γνωρίζουν κάποια ανάκαμψη, ενώ συγκρατούν την ανεργία, και από την άλλη υπάρχουν χώρες που γνωρίζουν ύφεση και διαρκώς αυξανόμενη ανεργία και κινδύνους ε, κοινωνικών ανταραχών. Το 2013 βρισκόμαστε στο τρίτο ευρωπαϊκό εξάμεινο, με ένα κύκλο για καλύτερο συντονισμό σε δημόσιονομικέ πολιτικέ των κρατών μελών, με τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής και τι κοινωνικέ μεταρρυθμίσει που απαιτούνται από τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να παρουσιάσω τι προτεραιότητε λοιπόν για τι κοινωνικέ αυτέ πολιτικέ στην όλη διαδικασία όπω έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο δεύτερο μέρο τη ομιλία μου θα ήθελα να τονίσω τη σημασία των πολιτικών αυτών και τη σημασία του συντονισμού από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για τις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές συνοχές και να δούμε ποια είναι τα δικαιβεύματα σήμερα όταν μιλούμε για την Δημοσιονομική και Οικονομική Ένωση και την κοινωνική της διάσταση. Θα ήθελα τώρα να σταθώ στην ετήσια έκθεση, ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη που δημοσιεύεται στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, όπως δημοσιεύτηκε τον Εύρο το 2012 ή το Δεκέμβριο. Ε, εδώ καθορίστηκαν προτεραιότητες για το 2013. Η έκθεση αυτή ορίζει τις βασικές προτεραιότητες για τις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές και στηρίζεται και από το σχέδιο της κοινή έκθεσης για την ε, ανα, ανάπτυξη, η οποία υιοθετείται ταυτόχρονα από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκθεση αυτή και η ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη έδειξαν μια ζωφερή εικόνα για την απασχόληση στην Ευρώπη. Με ένα ποσοστό 10,7% για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά στην ενεργεια. Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση σε πολλά κράτη-μέλη είναι πραγματικά <clears throat> σε διαρκή υποβάθμιση και υπάρχει κοινωνική αναταραχή. Η ετήσια επισκόπηση για το 2012 ήδη απαιτούσε την ε, καταπολέμηση της ανεργίας ιδίως των νέων και των κοινωνικών ανισοτήτων λόγω της ύφεσης η απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές είναι ακόμη πιο έντονες προτεραιότητες για τον οικονομικό κύκλο που έχει ξεκινήσει φέτος. Οι προτεραιότητε είναι η εξή. Δημοσιονομική εξυγίαση που θα πρέπει να είναι φιλική προ την ανάπτυξη ακόμη περισσότερο από ό,τι πέρυσι. Ενώ ο ρόλο των πολιτικών ανάπτυξη και απασχόληση θα είναι καθοριστική σημασία. Πάλι με στόχο την ανάπτυξη. Σε αυτή την επισκόπηση έχουμε εντοπίσει επενδύσεις στις οποίες θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα με φιλική προς την ανάπτυξη στάση και με δημοσιονομική εξυγίανση, δηλαδή δαπάνες οι οποίες είναι καθοριστικές για να διαφυλάξουμε το δυναμικό μας για μελλοντική ανάπτυξη, όπως ό,τι αφορά τις υπηρεσίες για την απασχόληση, τις ενεργές ε, πολιτικές για την αγορά εργασία, την εκπαίδευση και τα τονίζω αυτά γιατί είναι νέα στοιχεία καθώς και το ε, σύστημα της εγγύησης για την απασχόληση των νέων. Το Συμβούλιο των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΠΣΚΟ θα συζητήσει ακριβώς για την εγγύηση αυτή των νέων ένα πρόγραμμα που θα διασφαλίζει στους νέους κάτω των 25 σε τέσσερις μήνες αφού λάβουν πτυχίο ή μείνουν άνεργοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα διάστημα άσκησης ή μαθητεία και να έχουν κάποια θέση εργασία αυτό. Θα στηριχθεί παρόλο που δεν θα χρηματοδοτηθεί πλήρω από του δημοσιονομικού πόρου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια εμβληματική πρωτοβουλία, η οποία αποτελεί προτεραιότητα και για την νέα Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου. Επίσης σημαντικό είναι να τονιστεί ότι η δημοσιονομική ευθυγράμμιση θα πρέπει, και προσαρμογή θα πρέπει να διασφαλίσει κοινωνικά δίκτυα ασφαλείας όπως τον εξοχρονισμό των κοινωνικών ε, συστημάτων διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα, την καταλληλότητα και τη βιωσιμότητά τους. στα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλάβουν καλύτερα την έννοια των κοινωνικών επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ σύντομα θα εγκρίνει ένα πακέτο μέτρων για κοινωνικές επενδύσεις με ανάλυση και πρωτοβουλίες στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών, προκειμένου να γίνουν αυτές αποτελεσματικότερες και να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθειά τους να πετύχουν κάποιους τελικούς στόχους. Ο ρόλο των πολιτικών απασχόληση και των κοινωνικών πολιτικών είναι ζωτική σημασία για να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε τη κρίση. Να τονίσω κάποιε επιπλέον προτεραιότητε στου τομεί αυτού. Πρέπει να στηρίξουμε το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των οικονομιών μας. Ιδίω σε τρει τομεί που γοργά εξελίσσονται και ήδη είχαν εντοπιστεί πέρσι στο, στη δέσμη μέτρων για την απασχόληση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τομεί αυτή είναι η πράσινη οικονομία, όπω ονομάζεται, ο τομέα τη υγεία και των υπηρεσιών και ο τομέα ICT, υπεκινηνών και πληροφορική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν σφαιρικά μέτρα οι επενδύσει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδίω αυτού του γοργά εξελισσόμενου τομεί, είναι καθοριστική συνιστόσα, καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό θα πρέπει να αντικατοπριστεί σε όλε τι μελλοντικέ συζητήσει επίση για την ανταγωνιστικότητα τη οικονομία γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, είναι σημαντικό να πετύχουμε να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα και την δυναμικότητα των αγορών απασχόληση με ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις, ώστε οι αγορέ απασχόληση των κρατών μελών να γίνουν πιο ισόρροπες και περισσότερο συμμετοχικές και να προχωρήσουμε σε μια ευρωπαϊκότερη αγορά εργασίας. Τα μέσα για να στηρίξουμε την κινητικότητα των εργαζομένων παίζουν εδώ καθοριστικό ρόλο και η προτινόμενη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων για την αγορά απασχόληση των κρατών μελών θα πρέπει να βασίζονται στη συνεργασία με κοινωνικού εταίρου. Επίση, σημαντικό είναι οι φορολογικέ πολιτικέ να προσαρμοστούν στι απαιτήσει των καιρών. Το ίδιο και για του μισθού. Δεν θα πρέπει όμως να είναι πολύ μεγάλο το βάρος των ε, φόρων. Η εργασία που θα συσχετιστεί με σωστό τρόπο και με την φορολογία είναι προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό έχει γίνει, ε, αυτή η έμφαση έχει δοθεί και στα τρία ευρωπαϊκά εξάμεινα τώρα. Έπειτα έχει γίνει πιο οι έχουν γίνει πιο διορθωτικές ανάγκες της απασχόλησης. Ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 11 εκατομμύρια έχουν παραμείνει άνεργοι για περισσότερο από ένα χρόνο, οπότε πρέπει να δοθεί ειδική έμφαση στην αντιμετώπιση τη μακροχρόνια ανεργία. Και ταυτόχρονα να δούμε την ανεργία των νέων ω προτεραιότητα. Τέταρτο, θα πρέπει να δούμε κάποια βασικά δίκτυα ασφαλεία όπω τα ανέφερα. Αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Ξέρουμε ότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ μεταξύ των κρατών μελών ω προ την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών του συστημάτων. Υπάρχει περιθώριο για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των δημοσίων δαπανών ώστε τα κοινωνικά συστήματα προστασία να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά να υπάρξει μεγαλύτερη κοινωνική συμμετοχή και συμπερίληψη και να αποφευθεί ο αποκλεισμό. Η ενεργή συμμετοχή των ε, ενώσεων τη κοινωνία των πολιτών είναι κέρια σημασία για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών σε αυτόν τον τομέα, αλλά και για την ε, αποτίμηση, την αξιολόγηση. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για να τονίσουμε αυτή τη σημασία αυτού του θέματο, είναι η ένταξη των Ρωμά όπου έχει δημιουργηθεί στρατηγική πλαίσιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υλοποιεί χέρι με χέρι με τα κράτη-μέλη και τις ενώσεις ενδιαφερομένων ώστε να επιτευχθεί πρόοδος. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα θέμα για το οποίο μίλησε ήδη ο Αντιπρόεδρος, τις σημαντικές προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επανασχεδιάσει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Αυτό κατά την άποψή μου είναι θεμελιώδου σημασία με συστημικές απαιτήσει ώστε να ξεπεράσουμε τις οικονομικές, δημοσιονομικές, κοινωνικές και πολλές φορές και πολιτικές διαστάσεις της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Δεκέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ε, διατήρησα την εντολή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει μέσα και έναν οδικό χάρτη για, την για τον εξάντη συντονισμό των δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, για συμβάσεις αποτελεσματικότητας για την απασχόληση και την ανάπτυξη και μηχανισμούς αλληλεγγύης, προκειμένου να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Συμβόλιο επίσης έδωσε εντολή και στους δύο Προέδρους να διατηρήσουν μέτρα ώστε να διαφυλαχθεί και η κοινωνική διάσταση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού διαλόγου. Νομίζω υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα για να διατηρηθεί αυτή η κοινωνική διάσταση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση που θα πρέπει να προωθηθεί χωρί περαιτέρω καθυστερήσει. Ήδη χθε ε, στην διάσκεψη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αναφέρθηκε και από τον κύριο Ρεν παρουσίασα κάποιε ιδέε και θα ήθελα να αναφέρω κάποια στοιχεία. Νομίζω οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να τις δούμε πολύ σοβαρά. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιληφθούν ότι είναι αλληλοεξαρτώμενα και θα πρέπει να συνεργαστούν και καλύτερα προκειμένου να ξεφύγουμε από την κρίση. Στην ερχόμενη περίοδο θα πρέπει να οργανώσουμε ταυτόχρονη κινητοποίηση και, της δημοσιο... και του δημοσιονομικού συντονισμού και των δυνατοτήτων αλληλεγγύης για το ευρωπαϊκό αρχιτεκτόνημα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή σας και περιμένω την συνέχεια της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε και εμείς και περνάμε κατευθείαν στη συζήτηση. Αυτή τη στιγμή έχω 20 ερωτήσεις. 45 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι να δώσουν οι επίτροποι τις απαντήσεις τους. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Φρε... Φρέντο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, ε, καθότι έχετε πολλούς ομιλητές στο κατάλογό σας. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την, ε, την ε, τη δημοκρατική νομιμότητα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας στα εθνικά κοινοβούλια ε, σχετικά με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Δεν θα πρέπει να τους δώσουμε την εντύπωση ότι είναι αποκομμένα από την Ένωση. Βέβαια, κινούμαστε πάνω στα όρια και ξέρουμε ότι καταπατούμε το ιερό έδαφος των εθνικών κοινοβουλίων. Γι' αυτό θα πρέπει ε, να ε, είμαστε ευαίσθητοι ω προ το θέμα της εθνικής κυριαρχίας ε, και να εργαστούμε ώστε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ίσως θα πρέπει να βρούμε βέλτιστες πρακτικές ε, σχετικά με την διαδικασία διαβούλευση των Εθνικών Κοινοβουλίων κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό διότι είναι σημαντικό ε, να συμμετέχουν ε, ενεργά τα Εθνικά Κοινοβούλια της Ένωσης όσον αφορά την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ε, ε, είναι σημαντικό να έχουμε διαδικασία εξάντε και όχι εξπόστε, εκ των προτέρων και όχι των υστέρων. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει οικοδόμηση δυναμικού στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια όσον αφορά το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε την δυνατότητα ύπαρξης ενός προγράμματος της Ένωσης ώστε να διασφαλίζουμε ότι κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο, μικρό ή μεγάλο, θα έχει το απαραίτητο δυναμικό για να ασχοληθεί με τα θέματα θέματα αυτά. Βέβαια, περνάμε δύσκολου καιρού και όπω είπε ο Επίτροπο ε, Όλη Ρεν πολύ σωστά και συμφωνώ με αυτό, ε, θα πρέπει να ε, επιδείξουμε αλληλεγγύη σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ. Ταυτόχρονα πρέπει να φροντίσουμε να διατηρηθεί το κοινωνικό μα μοντέλο. Και νομίζω ότι το στοιχείο κλειδί εδώ, και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση, είναι ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο κατανόησης, ε, παρότι ε, θα πρέπει να έχουμε ενιαίους στόχους, να έχουμε σαφείς στόχους, ότι υπάρχει, ε, υπάρχουν διάφορες οδοί, διάφοροι δρόμοι στις διάφορες χώρες. Η κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρέπει, για παράδειγμα, να φροντίσουμε για παράδειγμα, η δική μου χώρα είναι μικρή χώρα, ε, περιορισμένο έδαφος ε, και είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε πολύ περισσότερο, αλλά ε, επειδή δεν δεν έχουμε πρόβλημα με τα ταξίδια, συχνά ε, έχουμε πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε η ε, οδηγία περί ε, χρόνου εργασίας δεν εφαρμόζεται πολύ εύκολα στη χώρα μας. Το μήνυμα που νομίζω ότι πρέπει να βγει από τη συνάντηση αυτή είναι ότι τα εθνικά κοινοβούλια συμμετέχουν στην προσπάθεια διατήρησης του ευρωπαϊκού μοντέλου, όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά, διότι το ένα δεν υπάρχει χωρίς το άλλο. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλίπ Μαρινή. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η παρούσα συνεδρίαση των εθνικών βουλευτών είναι δημοκρατικό άλοθη, άραγε ή ευκολόγιο κατάλογος καλών προθέσεων. Τόλμησα να αναρωτηθώ ε, κατά τη διάρκεια των δύο προηγουμένων συνεδριάσεων Νομίζω ότι τα πράγματα λίγο έχουν βελτιωθεί και προοδεύσει. Διότι έχουμε θέματα συγκεκριμένα, τα οποία έχουμε μοιράσει σε ε, συνεδριάσεις εργασίας. Έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, λέγω, διότι εάν δεν απατώμε, εκπροσωπείται και η Γερμανική Βουλή. Και δεν μπορώ να φανταστώ πως μια τέτοιου είδους συνεδρίαση Ευρωπαίων Εθνικών Βουλευτών θα ήταν ενδιαφέρουσα απουσία των Γερμανών Βουλευτών. Βέβαια, τούτων λεχθέντων απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. Έχουμε πρώτα απ' όλα τα προβλήματα με το ευρώ που ε, είναι και η πηγή των συνεδριάσεων μας. Ε, χάρη στο σύμφωνο ε, σταθερότητας ε, ε, έχουμε πιο μεγάλη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων εθνικών προϋπολογισμών και την εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των προγραμμάτων, ε, προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλησης κάθε χώρας. Ποια θα ήταν η δική μου ευχή. Στις επόμενες συνεδριάσεις να μπορέσουμε να κάνουμε μία διάκριση ε, στις συνόδους εργασίας μεταξύ των θεμάτων που συνδέονται απολύτως με τη σύγκληση ε, στην Ευρωζώνη αφενός και αφετέρου τα θέματα γενικότερης φύσεως τα οριζόντια εγκάρσια λεγόμενα που αφορούν ε, και τις 27 χώρες μέλη. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι για τις επόμενες συνεδριάσεις θα ήταν θεμητό και σκόπιμο να υπάρχει μια ε, προκατακτική ομάδα που να απαρτίζεται από εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων και ε, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορούν να προτείνουν τα θέματα εργασίας. Εάν θέλουμε πραγματικά να συμμετέχει με δημοκρατικό τρόπο ο κάθε βουλευτής που είναι πιο κοντά στους εκλογείς στις χώρες μας. Η επιθυμία είναι να μην επιβάλλεται το πρόγραμμα άνωθεν, αλλά ε, είναι απολύτως απαραίτητη να υπάρχει μια προεργασία συλλογική και σιγά σιγά να μπορέσει να αναδυθεί, να γεννηθεί κάτι το οποίο να μην εξυπηρετεί ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο, αλλά να είναι μοχλός όσο και φορέας πιο μεγάλης και πιο θεμητής και αποτελεσματικής συμμετοχής των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, στη μεγάλη ε, αυτή υπόθεση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας, ε, για την ε, ενίσχυση και εντατικοποίηση της συνεργασίας. Η κυρία Ποδηματά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον Ολυρέν και τον Επίτροπο Άντορς για τις παρεμβάσεις τους. Να ξεκινήσουμε από τα σημεία που συμφωνούμε γιατί υπάρχουν σημεία που συμφωνούμε ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σημαντικά. Συμφωνούμε, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιη ότι συμφωνούμε και στην συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων των Εθνικών Κοινοβουλίων με τις πέντε προτεραιότητες που έχουν οριστεί στην ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη. Μία δημοσιονομική προσαρμογή φιλική προς την ανάπτυξη, αποκατάσταση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, μεγένθηση και ανταγωνιστικότητα, αντιμετώπιση της ανεργίας και ένας αποτελεσματικός δημόσιος τομέας, δημόσιες υπηρεσίες. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς στην Ευρώπη που να διαφωνεί με αυτές τις προτεραιότητες. Το, μεγάλο στίχημα και το μεγάλο πρόβλημα ταυτοχρόνως είναι πώς θα μεταφέρουμε στην πράξη αυτές τις ε, προτεραιότητες στις οποίες συμφωνούμε, συμφωνούμε όλοι και όλες. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις και επ' αυτό νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε τη συζήτηση και να καταλήξουμε κάποια ερωτήματα προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το, η πρώτη προτεραιότητα, νομίζω, ε, είναι να σταματήσει αυτή η αλληλομετάθεση ευθυνών ως προς τις αιτίες της κρίσης. Βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα μια κατάσταση όπου πολλές εθνικές κυβερνήσεις μετέθεταν στο ευρωπαϊκό επίπεδο τις ευθύνες και αντιστοίχως από το ευρωπαϊκό επίπεδο υπήρχε μια στοχοποίηση στο εθνικό επίπεδο, ευθύνε στο εθνικό επίπεδο. Πρέπει να αναγνωρίσουμε νομίζω με γενναιότητα και ειλικρίνεια ότι υπήρξαν για αυτή την κρίση σοβαρές ευθύνε θεσμικές και πολιτικές και στο ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε θεσμικές και πολιτικές επάρκειες και στο εθνικό επίπεδο υπήρξαν λάθη και παραλήψεις σορευμένα από κρατημέλη που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Άρα να αναγνωρίσει ο καθένας τις ευθύνες του με γενναιότητα και ειλικρίνεια για να μπορέσουμε να πάμε παραπέρα. Το δεύτερο, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, και ε, αγαπητέ Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η πολύ σωστή προτεραιότητα για μια δημοσιονομική προσαρμογή φιλική ε, προς την ανάπτυξη. Ε, αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι όταν τα χρονοδιαγράμματα ε, δημοσιονομικής προσαρμογής εμφανώς ε, δεν βγαίνουν, θα πρέπει να έχουμε την ευελιξία να τα αναπροσαρμόζουμε. Και είναι σωστό αυτό που είπατε, αγαπητέ Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Υπάρχει αυτή η ακαδημαϊκή συζήτηση για την επίπτωση του δημόσιου χρέους όταν ξεπερνάει ένα επίπεδο στην ανάπτυξη, αλλά υπάρχει και μία άλλη συζήτηση σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δυστυχώς όχι τόσο πολύ στην Ευρώπη, κυρίως στο πλαίσιο άλλων οργανισμών, για την επίπτωση μιας απότομης δημοσιονομικής προσαρμογής στην ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν και τα δύο να τα δούμε για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε αποτελεσματικές πολιτικές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος από την Πολωνία. Ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, περιλαμβάνει κάποια θετικά αποτελέσματα, μεταξύ των άλλων ότι ε, θα έχουμε καλύτερη ε, οικονομική συνοχή. Επίσης, δημιουργούμε κίνητρα για μια μεγάλη συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά, την ανάπτυξη της οικονομίας δηλαδή, στα κράτη-μέλη αλλά η διαδικασία αυτή καθ' αυτή εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σημαίνει ότι ο διάλογος γίνεται κυρίως ανάμεσα στην Κομισιόν και τεχνικά Κράτη. Τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια παίζουν δεύτερο βιολί και δεν μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και έτσι είναι δύσκολο να μεσολαβούμε ανάμεσα στην ευρωπαϊκή πολιτική και τους πολίτες, διότι έχουμε ε, περιορισμένη δυνατότητα να την επηρεάσουμε. Υπάρχει και το άλλο θέμα του ε, ελέγχου της ε, διαδικασίας σε εθνικό, σε εθνικό επίπεδο, αλλά ε, και πάλι πρόκειται για διαδικασία που διεξάγεται ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στην Κομισιόν. Θα ήθελα ένα πράγμα να πω όσον αφορά την Κομισιόν. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερες διαδικασίες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα συζήτησης μεταξύ των κυβερνήσεων και των εθνικών ε, κοινοβουλίων όσον αφορά τα προγράμματα μεταρρύθμισης, ώστε να μην λαμβάνουμε απλά γνώση ε, ήδη λιμένων αποφάσεων. Δεύτερον, ο διάλογος αυτός περιλαμβάνει κάποιες ε, φάσεις στη συζήτηση, ε, κατά την οποία θα πρέπει να προετοιμάζουμε το πρόγραμμα μεταρρύθμισης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Ντανιέλ Ορουά. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρου τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την πρόσκληση που μα επιτρέπει να ανταλλάξουμε απόψει μεταξύ εκπροσώπων όλων των πολιτών τη Ένωση. Η σημερινή συζήτηση εντάσσεται στο, ε, ε, έτος, στο Ευρωπαϊκό Έτο των Πολιτών. Ένα ζήτημα που φαίνεται πολύ τεχνικό, ωστόσο μέσω των δημοσιονομικών μα επιλογών θα ε, διακυβευτεί το μέλλον μα. Η, Προεδρ... η Ιρλανδική Προεδρία θα κάνει τις επιλογές για την ανάπτυξη, για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, η επιλογή της βιώσιμης απασχόλησης ως προτεραιότητα θα σημαίνει ότι η λιτότητα δεν σημαίνει ανάπτυξη. Η υπερβολική λιτότητα αποτελεί κίνδυνο για όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Η Ευρώπη δεν μπορεί ενώπιον των χωρών του Νότου να χρησιμοποιεί τις ελεύθερες αγορές, τη λιτότητα και τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Η δημοκρατική ευθύνη βασίζεται σε αυτή την αντιπροσώπευση στα διάφορα κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων σωμάτων εντό τη Ένωση και οι πολίτε θα πρέπει να μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτό στο άρθρο 13 τη συνθήκη, όπω υπογραμμίζεται θα αποτελέσει το εργαλείο συνεργασίας μεταξύ όλων των κοινοβουλίων στην ε, Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Προσπαθούμε να ε, εμπλέκουμε τους συναδέλφους μας μέσω συνεδριάσεων για την οργάνωση του προϋπολογισμού μας. Κάναμε ένα γύρο τραπέζης στον οποίο συμμετείχε ο κ. Λαμασούρ, η κ. Περβόνς Μπερέζ, οι αρμόδιοι υπουργοί, οι επίτροποι, οι βουλευτές. Ε, ήταν εξαιρετικά διαφωτιστικοί. Όσον αφορά την έκθεση του Κριστοφ που κάθε δίπλα μου εδώ η Εθνοσυνέλευση υιοθέτησε ομόφωνα ένα ψήφισμα για την ταχεία δημιουργία του, ε, δημοσι... Δημοσιδικού Συνεδρίου που θα αποτελέσει εξαιρετικό εργαλείο για τη συνεργασία των βουλευτών για τα οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα που επηρεάζουν τόσο πολύ τους ανθρώπους. Θα ήταν πολύ καλό να μπορούσαμε να βρούμε μαζί μια κοινή μέθοδο που θα επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους αντιπροσώπους να συναποφασίζουν με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Έτσι θα μπορούσαμε να φύγουμε από τη σημερινή αντιπαράθεση που έχει ως αποτέλεσμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητά ε, μόνο ως συμβουλευτικό όργανο για τα δημοσιονομικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται, να βρουν την κατάλληλη μέθοδο συνεργασίας μεταξύ τους μέσω μια τέτοια συνόδου, να είμαστε πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί, όχι μόνο για τα δημοσιονομικά θέματα, αλλά και για όλα τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα επίσης. Να είμαστε αλληλέγγυοι για όλα τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος ε, Ταΐτης από τη Λιθουανία, παρακαλώ. Ε, Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όντως, είναι γεγονός ότι η σημερινή Ευρώπη δεν είναι Ευρώπη που οραματιστήκαμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, οικονομική κρίση, ασχολούμαστε αποκλειστικά με θέματα δημοσιονομικά και πολύ συχνά ξεχνούμε θέματα πιο πνευματικά ε, των κοινών μας αξιών. Το είπατε κι εσείς, ε, το είπε και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου. Κατά πολέμηση, λέμε, της ανεργία των νέων χρειάζεται μεγαλύτερη απασχόληση, να λαμβάνονται αποφάσεις, αλλά συγκεκριμένα δεν ακούμε κανένα μέτρο. Αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω. Δεύτερον, δεν λαμβάνονται τα μέτρα για να δημιουργηθούν καν οι ε, προϋποθέσεις. Αγαπητοί ε, παρισταμένοι, ε, συνεδριάζουμε σήμερα εδώ. Έχουμε ξανασυναντηθεί στο παρελθόν και στο μέλλον θα ξανασυναντηθούμε. Αποφάσεις παίρνουμε. Έχει κανένα αποτέλεσμα. Η ε, συνεδρίαση για την απασχόληση δεν κατάλαβα, δεν άκουσα τίποτα ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, τι γίνεται με τη φορολογία, με τους φόρους κατανάλωσης. Εγώ είμαι από τη Λιθουανία που συνορεύει με χώρες εκτός Ένωσης, που είναι η ε, Λευκορωσία και η Ρωσία. Έχουν ειδικούς φόρους κατανάλωσης ε, στα τσιγάρα και ε, στο ενόπνευμα, που είναι το 1 τρίτο το δικό μας και χάνουμε μέχρι και 5 δισεκατομμύρια ετησίως από εισόδημα φορολογικό όταν πηγαίνουν στις άλλες χώρες οι πολίτες μας. Ε, για την αγορά αυτών των προϊόντων. Λοιπόν, άλλο θέμα, ε, ενεργειακή ασφάλεια, ε, φοδιασμός. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε πολλούς ενεργειακούς πόρους και μέχρι τώρα δεν έχουμε μια κοινή προσπάθεια συντονισμού, συνεργασίας για να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Άλλο θέμα χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση της έρευνας και της επιστήμης στην Ευρώπη. Αυτά θα πρέπει να συζητάμε. Ωραίες κοινωνικές ε, ε, μορφές αλληλεγγύης ή η εγγύηση για τους νέους. Ωραία λόγια είναι, αλλά ε, στην πράξη τι κάνουμε για όλα αυτά. Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι κάθε νέος, και κάθε μεγαλύτερος οφείλει πρώτα απ' όλα να αναζητήσει ο ίδιο δουλειά και να φροντίσει για το εισόδημά του. Είπαμε, ε, θα ακολουθήσουν και άλλε συνεδριάσει, Ελπίζω όλα αυτά να γίνουν και πιο συγκεκριμένα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Η κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Επιτρόπους για όσα μόλις μας είπαν. Νομίζω κατέστη σαφές ότι η κατάσταση της ανεργίας είναι δραματική στην Ευρώπη. Όμω, εάν δεν δώσουμε πάλι δυναμικό χαρακτήρα στην οικονομία, δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και την ανεργία μακροπρόθεσμα. Ο κύριο Ρεν μα είπε με τρόπο πολύ σαφή ότι βλέπει ήδη θετικέ ενδείξει. Εγώ θα συμπλήρωνα λίγο αυτή την εικόνα διότι εάν αληθεύει ότι οι εξαγωγές αυξάνονται σε κάποιες χώρες, αυτό δεν αρκεί δεν αρκεί για να μπορέσει να μεγαλώσει και να αυξηθεί η οικονομία. Οι προβλέψεις πρέπει διαρκώς να αξιολογούνται εκ νέου και διαρκώς έχουμε και αρνητικές προβλέψεις. Υπάρχει μια διαρκή στάση προσήφεση και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά. Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως εντός της Ευρωζώνης υπάρχει πόλωση για να χρησιμοποιήσω τον όρο που χρησιμοποίησε και ο κύριος Άντορ επειδή υπάρχουν σοβαρές εσωτερικές αποκλίσεις στις χώρες με τα σοβαρότερα προβλήματα, η απώλεια του δυναμικού χαρακτήρα της οικονομίας δυσκολεύει και την δημοσιονομική ανάκαμψη. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε όχι μόνο τους πέντε στόχους της ετήσιας επισκόπησης για την ανάπτυξη επί των οποίων όλοι συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές ώστε να αντιμετωπίσουμε τη σοβαρότητα, την οξύτητα της κρίσης που και πάλι απειλεί τον κοινωνικό ιστό, την οικονομική συνοχή. Και συγκεκριμένα ερωτήματα τώρα. Δεν θα πρέπει τώρα να προσαρμοστούμε εκ νέου όχι απλώς στο στόχο της διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών, αλλά στο ρυθμό της προσαρμογής. Αυτόν δεν πρέπει να ξαναδούμε και να δούμε συγκεκριμένες συστάσεις με συγκεκριμένο ρυθμό για την προσαρμογή αυτή. Τα στοιχεία που θα αποτελέσουν μέτρα για την προσαρμογή δηλαδή της οικονομίας και έπειτα τι περιθώριο λιγμών έχουμε ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες επενδύσεις τι περιθώριο θα μας δώσει του χρόνου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να βρεθεί χώρος για τις επενδύσεις. Επενδύσεις απαραίτητες ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να λειτουργήσει μια στατική για την ανάκαμψη. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να δούμε στις προτάσεις της αιτήσεις επισκόπησης ε, ε, για την ανάπτυξη του 2013 μια πραγματική απόκριση στην οξύτατη κρίση η οποία συνεχίζει να ε, υπάρχει και να πλήττει την Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σερβές. Από το Ολλανδικό Εθνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ σήμερα, κύριε ο Ευχαριστώ το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διοργάνωση ε, είμαστε μέλη της ε, κάτω βουλής ε, του Ελλανδικού Κοινοβουλίου και χαιρόμαστε για την ευκαιρία που έχουμε να συναντηθούμε μαζί σας και συναδέλφους άλλων κρατών μελών για να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε πρώτα απ' όλα μια ευκαιρία αυτό να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές από τα κοινοβούλια μας για το πώς μπορούμε καλύτερα να αντιμετωπίσουμε τις νέες διαδικασίες και νέες μεθόδους του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ολλανδική Βουλή αποδίδει μεγάλη σημασία σε ένα σωστό διάλογο με τις κυβερνήσει μα για το ευρωπαϊκό εξάμεινο και αυτό απεικονίζεται και από το γεγονός ότι ορίσαμε και εισηγητή για το θέμα αυτό ε, που είναι πάρα πολύ σπάνιο στην Ολλανδική Βουλή. Χρειάζεται σε βάθος έλεγχος των κυβερνήσεών μας και αυτό είναι πρωταρχικός μας ρόλος. Ε, εγκαίρος ε, και με εύστοχο τρόπο, με πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες. Ε, θέλουμε διαφάνεια και ε, ε, θέλουμε επίσης τα περισσότερα έγγραφα και του Συμβουλίου, για να μην πούμε όλα, να είναι δημόσια και για μας και για το κοινό. Χαιρόμαστε για τον ενισχυμένο συντονισμό. και Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να βγει η Ευρώπη από την κρίση το ευρωπαϊκό εξάμεινο και η διαδικασία αυτή είναι σημαντικό στοιχείο ε, της όλης ε, σύσφυξης σχέσεων. Όπως γνωρίζετε ίσως στις κάτω χώρες γίνεται ζωηρή συζήτηση για την Ευρώπη αυτό τον καιρό. Ορισμένα κόμματα εκφράζουν περισσότερες επικρίσεις ε, για το μεγαλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενισχυμένο ευρωπαϊκό συντονισμό αυτών των πολιτικών στα κράτη-μέλη τι απαιτεί. Ο δημοκρατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο να οργανώνεται και να υπάρχει υποστήριξη ε, λαϊκή σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και η δική μα Βουλή αποδεί τόσο μεγάλη σημασία σε ένα ισχυρό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων σε όλα τα στάδια του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Ε, θα ήθελα να αναφέρω ένα άλλο ιδιαίτερο Ολλανδικό θέμα. Ε, το ε, Ολλανδικό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ προσιλωμένο στην αρχή της επικουρικότητας και αυτό κανονικά θα πρέπει να εφαρμόζεται και για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στις αρχές, στις πολιτικές, καταρχήν θα πρέπει να εκπονούνται αυτές σε επίπεδο κρατών μελών και οι συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις διάφορες χώρες θα πρέπει να παραμένουν σε γενικό επίπεδο ή μακροοικονομικό. Να στα κράτη-μέλη, στα κοινοβούλια και στις να έχουν πάντα το τελευταίο λόγο για ειδικέ επιλογές πολιτικής. Πρόεδρε, διασκέψεις αν αυτή μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη συζήτηση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα ισχυρό ρόλο για τα εθνικά κοινοβούλια και προσβλέπω στη συζήτηση ε, ε, μαζί σας σε επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Λόρδος Χάρισον από τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου. Κύριε Πρόεδρε, Έξι παρατηρήσεις. Πρώτο στον Όλιβερ, Όλιρεν. Ζητάμε από τους Γερμανούς ε, συναδέρφους ε, να ε, ελέγξουν τις εσωτερικές τους αγορές, αλλά πώς θα γίνει ο συντονισμός. Δεύτερον, με την ε, έκθεση ετήσιας ανάπτυξης, που είναι εξαιρετική ιδέα, πώς μπορούμε να μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι Ολλανδοί έχουν μόνο 9,7% ανεργία των νέων, ενώ υπάρχουν μέρη της Νότιας Ευρώπης που έχουν 50% ανεργία των νέων. Πώς θα μοιραστούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Ε, προς τον Επίτροπο Άντορ, τι εννοείτε όταν μιλάτε για ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Το σύνολο του προπολογισμού που διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή ε, δεν θα πρέπει να μετατραπεί σε ε, ε, προπολογισμό που να επικεντρώνεται στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει η Ευρώπη. Και όταν μιλάτε για προπολογισμό φιλικό προς την ανάπτυξη, πώς θα πετύχετε κάτι τέτοιο. Πώς μπορείτε να διασφαλίσετε η έρευνα και η ανάπτυξη, η καινοτομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βοήθεια προς μικρο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πραγματοποιηθεί. Και θα ήθελα να ρωτήσω τους τρεις προέδρους ε, το εξή σχετικά με τη γραφειοκρατία. Πολύ συχνά ακούμε ότι η υπερβολική ρύθμιση πνίγει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το όλο θέμα της ενιαίας αγοράς είναι να ε, μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Να γίνει κεράκι αντί για πυρκαγιά, αλλά ήρθε η ώρα η πολιτική να αντιμετωπίσουν ε, με αυτό το μάτι την ενιαία αγορά. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι ε, η Βουλή των Λόρδων που εδώ και χιλιάδες χρόνια ε, εκδίδει εκθέσεις όπως αυτήν για το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση. Και εμείς αλλάζουμε, έχουμε εφαρμόσει μέτρα λιτότητας Έχουμε εκπροσώπους από την Κύπρο, την ε, Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, ε, διότι θέλουμε να ακούσουμε την πραγματική τους φωνή. Εσείς ως ε, ευρωβουλευτές, τι κάνετε για να ακούσετε τις χιλιάδες φωνές που προσπαθούν να σας μιλήσουν. Και τέλος ένα ανέκδοτο. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο εξετάζει αν θα γίνει δημοψήφισμα στο αν θα παραμείνουμε ή όχι στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαβάστε παρακαλώ την ομιλία του Πρωθυπουργού, διότι έχει πολλά ε, καλά στοιχεία. Εδώ και πολλά χρόνια ήμασταν ε, οι γείτονε που κάναν φασαρία. Εγώ ήμουν πάντα Ευρωπαίο, θα είμαι πάντα Ευρωπαίο. Ε, πιο ταπεινή μου φιλοδοξία είναι να, της Ευρωπαϊκής, να είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να είμαι και η φωνή του, του πάρτι, να είμαι ο, πιο ζωηρό άνθρωπο στο πάρτι. Unser έχουμε ως σύνθημα ενωμένη στη διαφορετικότητα. Αυτό είναι το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό έχουμε ε, συνέλθει εδώ για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας και να λύσουμε από κοινού τα κοινά μας προβλήματα. Η κυρία ε, ε, Βετίνα Κούτλα από τη Γερμανία. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, λέει η κυρία Κούτλα, χαιρόμαστε πάρα πολύ για την ευκαιρία που έχουμε ε, με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να προωθήσουμε την εξηγίαση των δημοσίων οικονομικών και των προπολογισμών και να κάνουμε προσπάθειες ε, για να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μεμονωμένων χωρών. Επίσης είναι ευπρόσδεκτο και το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Προτάσετε λίγο χρονικά κατά τη διάρκεια του έτους αυτό τα εθνικά σχέδια στο μέλλον θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού στα διάφορα κράτη-μέλη. Και σκοπός είναι τώρα να φροντίσουμε όσο γίνεται αυτή η δημοσιονομική διαδικασία να μπορεί να βαίνει απρόσκοπτα και χωρίς ε, αναταραχές. Είναι μεγάλες όμως και οι προκλήσεις. Μόλις ακούσαμε ότι η Μεγάλη Βρετανία σκέφτεται να κάνει ενδεχομένως ένα δημοψήφισμα θα πρέπει αυτές οι επιφυλάξεις να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να έχουμε οπωσδήποτε ε, επίγνωση του τι στη εσωτερική αγορά στην Ευρώπη. Και πόσο θα αποδυναμωνόταν αυτή ε, αν φύγει η δεύτερη μεγαλύτερη εθνική οικονομία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια θα ήταν η θέση μας ανταγωνιστικά απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο. Και η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών και των προπολογισμών σε μια πολιτική που είναι φιλική προς την ανάπτυξη. Αυτή και πάλι η πολιτική ε, με τη σειρά της συνδέεται στενά με την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο οι προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κατά τόπους. Δεν επιτρέπεται να μην λαμβάνονται υπόψη τα τοπικά δεδομένα και ιδιαιτερότητες ορισμένων κλάδων της οικονομίας, για παράδειγμα, ή ε, κάποια δεδομένα της πολιτικής κατάστασης εκάστοτε τόπου διότι συχνά υπάρχει εναγκαιότητα να λαμβάνετε υπόψη ότι έχουμε κυβερνήσει συνεργασία και συνασπισμού που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη του διάφορου εταίρου. Τι προτείνει η Κομισιόν για τη Γερμανία, Να ε, καταργηθεί ε, ε, ο διαχωρισμός ο φορολογικός των συζύγων ή το επίδομα τέκνων. Μα αυτό είναι θέμα οικογενειακής πολιτικής, εθνικής. Δεν λύνει το πρόβλημα της εξυγίασης των δημοσίων οικονομικών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα δημόσια οικονομικά και στο τι επιβαρύνει τον προπολογισμό. Και αυτά είναι θέματα, α πούμε, τα προβλήματα τη κοινωνικής ασφάλισης, αγορά εργασίας, σύνταξη και ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Θα πρέπει να βρεθούμε, λοιπόν, σε μια κατάσταση να δούμε πώς θα συμμετέχει το κράτος σε αυτή τη χρηματοδότηση και πώς ε, το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου θα εφαρμόζεται. Αυτό το σχήμα θα πρέπει ε, να είναι ακόμα αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Ακόμα δεν υπάρχει απαραίτητη δημοκρατική νομιμότητα. Μα και γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει εδώ, ο Πρόεδρος, γιατί θα πρέπει να συνεννοηθούμε στο ποια μορφή θα λάβει αυτό. Τώρα έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Σε 7 λεπτά θα πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχω ακόμα 15 ομιλητέ. Σας παρακαλώ όσο γίνεται να τηρείτε το χρόνο σας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τραβήξω μια γραμμή σας παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι και να κάνετε ερωτήσεις. Κύριος Γιούκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, βρίσκομαι εδώ κύριε Επίτροπε. Το έγγραφο κλειδί είναι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για αυτό το Ευρωπαϊκό Εξάμενο στην ε, Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του παροντός Κοινοβουλίου δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά την ε, εκτίμηση αυτής της αιτήσης ανασκόπηση. Η δημοκρατική συζήτηση είναι πολύ σημαντική για αυτό το ζήτημα. Η δική μας ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, έχει δύο αντιρρήσει για την έκθεση που παρουσιάζεται. Η πρώτη σχετίζεται με την αξιολόγηση τη Κομισιόν όσον αφορά τον πολλαπλασιαστή. Όπως γνωρίζετε, το Δουνουτού που ανήκει στην ίδια τρόικα μέσα ε, αυξάνει τον πολλαπλασιαστή. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον είχατε υποτιμήσει την, ε, ε, τις επιπτώσεις υπέρ της ύφεσης των πολιτικών που προτείνετε εσείς. Η δεύτερη αιτία Όσον αφορά το ρυθμό του χρονοδιαγράμματος της ομοίωσης των ελλημάτων, έχουμε κάποια ερωτηματικά. Ο ρυθμός μείωσης των ελλημάτων που προτείνει η Κομισιόν, προτείνετε εσείς, για ορισμένες χώρες του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης είναι 1,5% μείωση του ελλήματος ενώ το six-pack μειώνει ε, επιβάλλει ε, μείωση του ελλήματος μόνο κατά 0,5% σήμερα βρισκόμαστε σε ύφαση εντός της Ευρωζώνης το διαρθρωτικό έλλειμμα που μας επιβάλλει μας επιβάλλεται σε ορισμένες χώρες θα ισορροπηθεί ήδη ε, στην Ιταλία νομίζω χάρη στις προσπάθειες και στη Γαλλία ε, θα υπάρχει δυνατότητα διαρθρωτικού ελλείμματος ε, σχεδόν μηδέν και κανονικού ελλείμματος άνω του 3%. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους ύφεση. θα δεχθείτε να αναθεωρήσετε τις συστάσεις που κάνετε και να Ακολουθήστε το Sixpack, τη δεσμή 6 μέτρων που φαίνεται καταλληλότερο από τις σύστασεις που κάνετε εσείς ε, δεδομένων των τρεξών συνθήκων. Επίσης, ε, θα ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο Μαρίνη από την Γαλλική Γερουσία. Εγώ δεν είμαι αντίθετο του δημοκρατικού ελέγχου σε ευρωπαϊκή κλίμακα και στα κράτη-μέλη και του δημοκρατικού ελέγχου στα κράτη-μέλη. Είμαι υπέρ και των δύο. Γι' αυτό τον λόγο ζητάμε σε περίπτωση αλλαγή των συνθήκων να αποτελέσει νομοθετική ε, πράξη, η ετήσια ανασκόπηση, αλλά θα ήθελα να ε, μας πούν την αψίδα να ψηφίσω για τα εθνικά προγράμματα σταθερότητας. Ευχαριστώ κύριο Ρενέ Βανερ Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπορώ να είμαι πολύ σύντομος. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιτρόπους για ε, τη δέσμευσή τους. Θέλω να προσθέσω τα εξής δύο. Πρώτον, Ευρώπη των δύο ταχυτήτων είμαι υπέρθερμος υποστηρικτής αυτών των δύο ταχυτήτων. Μιλάμε για διαφορετικές Ευρώπες στην Ευρώπη. Και δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη à la carte κατ' επιλογή. Τότε να ξεχάσουμε όλες ε, τις συζητήσεις που κάνουμε στα Εθνικά Κοινοβούλια. Χρειάζεται λοιπόν συζήτηση για την Ευρώπη ταχυτήτων. Το δεύτερο. Ε, η Ευρώπη έχει πρόβλημα εικόνα και αυτή η εικόνα σχηματίζεται στα εθνικά κοινοβούλια για του λαού. Θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν και μεγαλύτερο ρόλο και μεγαλύτερη δέσμευση. Είναι αδιανόητο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο χωρίς να συμμετέχουν και να έχουν μεγάλο ρόλο πρωταγωνιστικό τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί πολλά στοιχεία έχουν να κάνουν με εθνικές αρμοδιότητες και εξουσίες. Αλλά η εικόνα λοιπόν που διαμορφώνεται για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ κακή. Και το λέγω εδώ αυτό διότι σε πολλές περιπτώσεις η Ευρώπη παρουσιάζεται ως μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι γραφειοκρατική, που είναι σπάταλη, που ασχολείται με πάρα πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε. Αυτό εν μέρη μπορεί να ισχύει, αλλά θα πρέπει να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα για την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο αγορά η Ευρώπη. Είναι πολύ περισσότερο και δεν είναι το πρόβλημα. Είναι μέρο τη λύση η Ευρώπη. Γι' αυτό ζητώ οπωσδήποτε να συζητήσουμε αυτό το θέμα και τη Ευρώπη των δύο ταχυτήτων και το να έχει στο μέλλον η Ευρώπη ίδιου πόρου. Έτσι ώστε να μην μπαίνουμε σε αυτή ε, τη διαδικασία και τον καυγά μεταξύ των καθαρών συνεισφορέων και των καθαρών αποδεκτών. Αυτό στρεβλώνει τη εικόνα τη Ευρώπη στου πολίτες. Και αν δούμε τα πραγματικά στοιχεία, πού αυξάνονται οι δαπάνες, στους εθνικούς προϋπολογισμούς, όχι στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, να είμαστε αυτοκριτικοί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει την αυτοκριτική του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις δαπάνες και τον τρόπο με τον οποίο αυτές ε, δίδονται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνετε ότι εγώ δεν χαίρομαι πολύ με τα ε, χειροκροτήματα. Ο κύριος Χρυσόγελος, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων εθνικών κοινοβουλίων. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να συμμετάσχουν και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών για αυτή τη συζήτηση συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Βέβαια, όταν μιλάμε για συντονισμό οικονομικών πολιτικών και δημοσιονομική εξυγίανση, πρέπει αυτές οι πολιτικές να είναι συμβατές με τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με τους στόχους Ευρώπη 2020 και κοινωνική συνοχής. Δεν μπορεί η δημοσιονομική εξυγίανση να καταστρέφει την κοινωνική συνοχή, να διαλύει την οικονομία και να αυξάνει σε, αυτή την σε αυτόν τον εκρηκτικό βαθμό την ανεργία. Είπε ο Επίτροπος Απασχόλησης ότι η δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει να προστατεύει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Πολύ σωστό. Όμως αυτό δεν είναι μέσα στις στρατηγικές δημοσιονομικής προσαρμογής σήμερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. Αντίθετα, καταστρέφεται το δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Είπε ο επίτροπο κ. Όλη Ρεν ότι βελτιώθηκε η ανταγωνιστικότητα τη ελληνική οικονομία. Αυτό δεν έγινε όμω με βάση την καινοτομία, την αναδιοργάνωση τη εργασία, την αποτελεσματική οργάνωση τη διοίκηση, αλλά έγινε με υπερβολική περικοπή των μισθών. Άρα δεν είναι βιώσιμη μακροχρόνια. Ποιοι είναι οι τομεί καινοτομία. Οι τομεί καινοτομία είναι η πράσινη οικονομία, η η τεχνολογία, η πληροφορική, όμως αυτά δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική που να συνδυάζεται με τους στόχους Ευρώπη 2020 όταν μιλάμε για δημοσιονομική εξυγίανση. Είναι αποτυχημένη αυτή η στρατηγική που εφαρμόζεται και θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία να προσαρμόζεται η στρατηγική στις πραγματικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί πολλέ φορέ ότι έγιναν λάθο εκτιμήσει για το δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι τα μέτρα λιτότητα και περικοπή να αυξάνουν το χρέο. Στην πραγματικότητα, εάν υπήρχε σταθερότητα τη οικονομία στο επίπεδο του 2011, θα, μειώνονταν το χρέο κατά 20%. Ενώ σήμερα η πολιτική που εφαρμόζεται αυξάνει το χρέο σε εκρηκτική διάσταση. Και βέβαια <clears throat> τα θέματα τη απασχόληση. Δεν μπορεί η κοινωνία να βλέπει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές εστιάζουν μόνο σε περιοριστικά μέτρα και δεν επιλύουν τα άλλα προβλήματα όπως είναι η απασχόληση, η κοινωνική συνοχή. Θέλουμε λοιπόν και δημοκρατικό έλεγχο αυτών των πολιτικών που σήμερα εφαρμόζονται και ισορροπημένες πολιτικές για την απασχόληση, την αναζωγόνηση της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή. Uh, Mr. Nikos Ευχαριστώ κύριος Νικολαίδης παρακαλώ. Cyprus. Από την Κύπρο. Thank you, President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κοινοβουλευτική εβδομάδα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι ε, ε, μια εκδήλωση της οποίας όλοι, όλοι καταλαβαίνουμε τη σημασία η κοινοβουλευτική συνεργασία ανάμεσα στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να ε, δημιουργήσει την απαραίτητη ορμή και τις συνέργειες ε, για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένωση αμφισβητείται. Ε, δεν είναι μυστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε βαθιά και πολλαπλή κρίση. Για να βρούμε τις σωστές λύσεις θα πρέπει πρώτα να βρούμε τις αιτίες του προβλήματος και Βέβαια δεν θα βρούμε τις σωστές αιτίες αν ε, κοιτάζουμε προς τη λάθος κατεύθυνση. Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά δημοσιονομικό, είναι ε, απλά ε, αριθμητική έκφραση του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι η οικονομική κρίση και ε, το ότι η οικονομία δεν κινείται. Τα προβλήματα αυτά είναι συστημικά και επιδονώνονται από την χρηματοπιστωτική κρίση στην οποία έχουμε οδηγηθεί λόγω της διεθνούς τραπεζικής κρίσης. Καταρχήν, λοιπόν, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά προβλήματα και δεύτερον, θα πρέπει να διατηρήσουμε ε, την πορεία μας ε, προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σημαντικό είναι να επιλέξουμε τις δράσεις μας με τρόπο ώστε να εξυπηρετούμε και τους δύο στόχους ταυτόχρονα. Δεν θα πρέπει όμως να χάσουμε την επαφή μας με τις βασικές ε, αξίες ε, και αρχές ε, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντικειμενικότητα, η αλληλεγγύη και επιδίωξη του κοινού καλού. Στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε προς την ολοκλήρωση με ισορροπημένα βήματα βήματα προς ολοκλήρωση της αγοράς που ακολουθήθηκε από ένα βήμα για την κοινωνική συνοχή. Ε, σήμερα όλο και περισσότερε χώρε αντιμετωπίζουν βαθιά οικονομικά προβλήματα. Ο τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει συλλογικά τι χώρε αυτέ ε, θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον των χωρών αυτών, αλλά και το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Ε, είναι λογικό ο βασικό στόχο ε, να είναι να υποστηρίξουμε τι ε, ασθενεί οικονομίε, προστατεύοντα τι ισχυρέ οικονομίε και την οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Οποιοδήποτε πρόγραμμα διάσωση που θα συμφωνηθεί ε, προς κάποια χώρα θα πρέπει για να είναι επιτυχές να λαμβάνει υπόψη τα, ε, ε, τα βασικά στοιχεία της οικονομίας που θα πρέπει να διασωθεί. Θα πρέπει λοιπόν να εξεταστούν όλες οι πτυχέ της οικονομίας αυτής με αντικειμενικό φυσικά τρόπο. Τα δημοσιονομικά προβλήματα, το σύστημα φορολογίας, ο τραπεζικό τομέας και θα, πρέπει να εξεταστούν και οποιασδήποτε στρεβλώσεις περιέχει ένα τέτοιο σύστημα. Ε, η, εξέταση αυτή θα πρέπει να γίνει ε, ε, με ευρύ τρόπο και ο Πρόεδρος διακόπτει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπάκης. Είναι σαφές ότι η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να διαμορφώνεται και να εφαρμόζεται αγνώντας τις κοινωνικές συνέπειες, τη δυναμική δηλαδή της απασχόλησης και της ενεργείας αντίστοιχα η ιστορία έχει αποδείξει ότι χωρί τη συνένεση τη κοινωνία, καμιά μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι επιτυχημένη και κανένα οικονομικό πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Είναι λοιπόν αναγκαίο αφενό να ενισχυθούν και να συμφιχτούν οι σχέσει εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω μέσο προαγωγή τη δημοκρατική νομιμοποίηση του εξαμήνου και αφετέρου επιβάλλεται οι δρομολογούμενε πολιτικέ να σχεδιάζονται με κοινωνική δικαιοσύνη και αναπτυξιακή πνοή η ιδέα υλοποίησή του να πραγματοποιείται πάντοτε σε συνθήκε κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση και με την ευκαιρία που βρίσκεται ο Αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Όλι Ρεν, και ο Επίτροπο κ. Σαντόρ, θα ήθελα να επισημάνω και να ρωτήσω με ποιο τρόπο διασφαλίζεται στην πράξη ότι τα διακονομικά πλάνα που υιοθετούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όχι μόνο δεν λειτουργούν σε βάρο τη κοινωνική συνοχή και τη απασχόληση, αλλά αντίθετα προάγουν τους στόχους της στρατηγικής 2020 για καταπολέμηση της ανεργίας και μείωση της φτώχειας τόσο άμεσα σήμερα όσο και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο ακόμα σε δύο συναδέλφους, γιατί ο Επίτροπος κύριος Άντορ πρέπει να αποχωρήσει λίγο. Ο κύριος Ρόσμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η ψηλή ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανησυχεί πάρα πολύ. Αλλά με ανησυχεί και πολύ και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε αυτές τις προκλήσεις που μας έχει φέρει η κρίση. Γιατί οι απαντήσεις είναι πάντα ίδιες. Η στρατηγική των τριών πυλώνων που βασίζεται βασικά σε εξυγίανση του, οικονο... Ε, του προ υπολογισμού, ανταγωνιστικότητα και διαρθρωτικά μέτρα. Αν δούμε την εξηγίαση του προπολογισμού θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε μια αποτελική λιτότητα με κάθε τίμημα σε μια κατάσταση όπου κανονικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανάπτυξη για να επιτύχουμε την απασχόληση. Η Ευρωζώνη είναι σε ύφαση, οπότε δεν είναι και απορία άξιο που αυξάνονται οι κριτικές για την πολιτική του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερο. Και πρόσφατα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει νέες ε, εκτιμήσεις ε, για τον πολλαπλασιαστή ο κύριος Ολιβιέ Μπλανσάρ, επικεφαλής των οικονομολόγων και πολύ σημαντική είναι η κριτική της κυρίας Λαγκάρτ και πρόσφατα είδαμε ότι η πολιτική τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεωρείται με πολύ κριτικό μάτι γιατί δεν μας φέρνει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αντίθετο, ε, βυθίζεται πιο βαθιά στην κρίση η Ευρώπη είναι μακρά στασιμότητα με διατήρηση υψηλής ανεργίας και όχι καταπολέμηση της ανεργίας. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι μια συστημική απάντηση σε μια συστημική κρίση. Ε, αυτή την απάντηση δεν την έχουμε. Ακόμα και αν προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και κάπως να διορθώσουμε τα πράγματα, να ε, διαμορφώσουμε πιο ισχυρά τον οικονομικό χώρο, αλλά παρακολουθώ και διαπιστώνω ότι η στρατηγική μας ουσιαστικά ποια είναι. Περικοπές μισθού στην περιφέρεια, ε, στα περιφερειακά κράτη, εσωτερική υποτίμηση. Μέχρι πού θα γίνει λοιπόν αυτή η εσωτερική υποτίμηση, πού θα φτάσει. Πόσο καιρό θέλουμε ακόμα να παραμένουμε θεατές ε, ε, για το πώς υπάρχουν ε, επεμβάσεις στα θέματα των συλλογικών συμβάσεων και στα μισολογικά. Ο Διεθνής Οργανισμός Απασχόλησης αντιδρά ήδη. Μα πώς θα δημιουργηθεί έτσι η απασχόληση και θα καταπολεμηθεί η ανεργία. Συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Τι απέγινε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που δημιουργήθηκε πέρσι το καλοκαίρι. Μέχρι τώρα είναι κενό γράμμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πλάνκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάρας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπη για τις παρουσίες σας ως μέλος του Εθνικού Κοινοβουλίου και παρατηρητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους μας τους συναδέλφους εδώ που ήδη επικύρωσαν την συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας και αναμένουμε τις πέντε προχωμένες επικυρώσεις που ελπίζουμε να γίνουν αγερά. Μια σύντομη ενημέρωση και ένα σημείο για την Κροατία που έχει ξεκινήσει έναν εντατικό διάλογο με την Κομισιόν για να συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο πριν ολοκληρωθεί η προσχώρηση. Οι στόχοι του ετήσου προγράμματος ανάπτυξης αποτελούν κομμάτι του μελλοντικού οικονομικού προγράμματος και του προγράμματος σύγκληση ε, που θα υποβληθεί στην Κομισιόν μέσα στους επόμενους μήνες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τις απόψεις της Επιτροπής όσον αφορά το πώς η επίσημη συμμετοχή της Κροατίας στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πρόκειται να υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ ο, Επίτροπος κ. Σαντόρ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Θα αναγκαστώ να είμαι πολύ σύντομος. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πλούσια η συζήτησή μας. Βέβαια κράτησε λίγο παραπάνω από ό,τι περιμέναμε, οπότε θα πρέπει να συνοψίσω τις απαντήσεις μου. Πάντως, κάποιες από τις βασικές παρατηρήσεις που έγιναν στην όλη συζήτηση, ιδίω ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Νομίζω ότι ήταν βάσιμες οι ανησυχίες που εκφράσατε οι περισσότεροι από εσάς, ιδίω από τις περισσότερο περιφερειακές ε, χώρες και μάλιστα όσες ανήκουν στην Ευρωζώνη. Να υπογραμμίσω ότι κάποιες φορές υπάρχει εδώ μια αντίφαση στις αναλύσεις που γίνονται. Από τη μια δεν μπορούμε να επιμένουμε στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και από την άλλη να επικρίνουμε την βασική νομοθεσία σε αυτό το τομέα, όπως την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Η οδηγία αυτή είναι σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, αναπόσπαστο στοιχείο. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, να καταπολεμήσουμε την άνηση μεταχείριση, το κοινωνικό ντάμπινγκ και αυτή ακριβώς είναι η δουλειά της εφηούς νομοθεσίας. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της νομοθεσίας εφόσον ε, χρειάζεται μάλιστα να ευθυγραμμίζουμε, γιατί δεν υπάρχει ποτέ ένα μέγεθος για όλα και μία λύση για όλες τις περιπτώσεις, αλλά αυτό είναι το σοβαρότερο έργο που έχουμε να επιτελέσουμε. Να τονίσω εδώ ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χώρο αυτό δεν θα αποτελούσε ποτέ φραγμό στην οικονομική ανάπτυξη η ίδια η αντίληψη της, ε, η οδηγία ή ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να στραγγαλίζει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ένας επικίνδυνος μύθος. Θα πρέπει εδώ να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους τους μύθους, ε, τις ιδεολειψίες με πραγματικά επιχειρήματα. Η ο κανονισμος της ευρωπαικης ενωσης θα μπορουσε να στραγγαλιζει την ευρωπαικη νομοθεσια ειναι ενας επικινδυνος μυθος θα πρεπει εδω να καταπολεμησουμε αυτου του ειδους τους μυθους της ιδεολειψιας με πραγματικα επιχειρηματα η υφεση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οφείλεται σε διαφορετικά αίτια και μάλιστα σε κάποιε περιπτώσει η ανάκαμψη έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο καιρό. Τώρα για τα ευρωπαϊκά δημοσιονομικά εργαλεία και μέσα. Εδώ μπορούν να διαδραματίσουν ένα θετικό ρόλο, ακόμη και μέσω των διαρθωτικών ταμείων, προκειμένου να αποκριθούμε στην κρίση με τρόπο ε, ε, ευελιξία, με ευέλικτο τρόπο. Πολλά κράτη-μέλη προσαρμόζουν τα προγράμματα μεταρρυθμίσεών τους ώστε να ευνοήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασία, να ευνοήσουν την απασχόληση. Γι' αυτό κάποιε φορέ για τι χώρε μνημονίων έχουμε προβλέψει διαφορετικά ποσοστά συγχρηματοδότηση, ώστε να ε, επιτρέψουμε να δημιουργηθούν οι κατάλληλε ε, συνθήκε. Επίση, η Επιτροπή πρόσφατα διαδραμάτισε ενεργό ρόλο με την αποδέσμευση κονδυλίων ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων στα οκτω κράτη-μέλη που έχουν πληγεί σοβαρότερα και έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά. Εδώ να τονίσουμε τη δυνατότητα μεταφοράς των βέλτιστων πρακτικών σε χώρες που τις χρειάζονται και έχουν προβλήματα. Πολλά ερωτηματικά έχουν τεθεί σχετικά. Πάντως, ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι η εγγύηση για τους νέους. Έχει λειτουργήσει σε χώρες όπως η Αυστρία και η Φινλανδία. Έχουμε μάλιστα αναπτύξει μια τέτοια έννοια στη δέσμη μέτρων για τους νέους, προσπαθώντας αυτές τις βέλτικες πρακτικές να τις ε, εφαρμόσουμε σωστά και αλλού. Γι' αυτό οι σχετικές συζητήσεις του Συμβούλου είναι τόσο σημαντικές και γι' αυτό είναι σημαντικό όλα αυτά να μεταφερθούν στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας ε, και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω τα εργαλεία αυτά, τα μέσα αυτά έχουν προστιθέμενη αξία. Μιλάμε για κονδύλια για τις ε, επενδύσεις. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από εθνικούς πόρους, από έλεγχο και αναλύσεις του κινδύνου βεβαίως την παρακολούθηση του κατά πόσον δαπανώνται νόμιμα τα κονδύλια αυτά και βεβαίω του συντονισμού ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικών περιφερειακών επιπέδων, ώστε να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα για την διαδικασία προσαρμογής και τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων, αυτά όλα είναι περίπλοκα βέβαια, αλλά όταν μιλάμε για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να επιτρέψουμε την προετοιμασία των προγραμμάτων αυτών και την συμμετοχή των εθνικών παράγοντων συγκεκριμένα, των κοινωνικών εταίρων για τι συνταξιδοτικέ μεταρρυθμίσει λόγου χάρη. Μαζί με τον κύριο Ρεν και τον κύριο Μπαρνιέ το 2010 δημοσιεύσαμε μια πράσινη βίβλο η οποία ακολουθήθηκε και από μια λευκή βίβλο και ξεκίνησαν συζητήσεις με τους εθνικούς φορείς για τα έγγραφα αυτά. Έτσι χαράξαμε το δρόμο για να φτάσουμε στην ανάλυση των συνταξιωτικών συστήματων στις αιτήσει επισκοπήσεις της ανάπτυξης ώστε να οδηγηθούμε σε χειροπιαστές συγκεκριμένες συστάσεις και ήδη αυτό από τα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά εξάμεινα. Προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο σε επίπεδο κοινοτικό με διαβουλεύσεις αλλά και διάλογο με τους πλέον ενδιαφερόμενους. Πριν φτάσουμε στις συγκεκριμένες όπως έλεγα συστάσεις. Εγώ ο ίδιο συμμετείχα σε συζητήσει σε εθνικά κοινοβούλια όπω τη Γερμανική Bundestag, το Ιταλικό Κοινοβούλιο, την Πορτογαλική Βουλή, προηγουμένω στη Φιλανδία, στην Ελλάδα και δεχόμαστε και προσκλήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό για μας είναι άκρο σημαντικό, διότι επίσης δείχνει ότι η επισκόπηση για την ανάπτυξη και οι συστάσεις δεν στοχεύουν απλώς στις χώρες οι οποίες έχουν οικονομικές δυσχέρειες αλλά έχουν, ε, συμπεριέχουν και περιέχουν σημαντικές προτάσεις για όλους και για χώρες που λειτουργούν πιο εύρυθμα, όπως η Γερμανία θέλουμε να γίνει αντιληπτό ότι είναι πολύ σημαντική η αρμοδιότητα της ε, πολιτικής απασχόλησης να αντιμετωπίσει τις ανισορροπίες, τις ανισότητες, την έλλειψη ισότητας μεταξύ των φύλων, ε, την διόρθωση των ελάχιστων μισθών στην αγορά εργασίας. Προσπαθούμε λοιπόν να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σφαιρικοί στην αντιμετώπιση μας, να επιτρέπουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και ελπίζουμε ότι η μέθοδος αυτή που έχουμε ξεκινήσει να χρησιμοποιούμε θα μας ε, οδηγήσει στα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα και την ικανοποίηση όλων των συμμετεχόντων. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστούμε πολύ κύριε Άντορ. Έξι ομιλητές έχουμε, αλλά θα δώσω το λόγο μόνο σε δύο. Οι άλλοι θα πρέπει να μιλήσουν στις διάφορες επιτροπές, διότι πρέπει να ακούσουμε τις απαντήσεις του Επιτρόπου ΡΕΝ και για τις ε, συναντήσεις που θα έχουμε το απόγευμα. Αλλά θα δώσω το λόγο σε δύο μιλητές ε, από χώρες ε, από τις οποίες δεν ακούσαμε κανέναν μέχρι τώρα. Από τη Φιλανδία καταρχήν εκτός μικροφώνου. please. Κυρία Κούμπουλα Νάτρη από τη Φιλανδία. Έχω τρεις παρατηρήσεις από την ε, φιλανδική άποψη. Αναμένουμε το εξάμεινο να εξετάσει και τις νέες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στους ε, προϋπολογισμούς. Από θεσμική άποψη θεωρώ ότι καμία σύνοδος ε, δεν μπορεί να είναι σε θέση να παρέχει δημοκρατική εξέταση, η νομιμότητα. Είναι σαφές αυτό. Ακόμα και αν δύναμη του νέου άρθρου 13 μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό φόρουμ, χρειαζόμαστε ένα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε εξουσία σε εθνικά κοινοβούλια, έχουμε εξουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το λιγότερο που μπορεί να μένουν οι άνθρωποι είναι το να τα αναμίξουμε και να τα κάνουμε ακόμα λιγότερο σαφή. Πιστεύω ότι όλα τα κοινοβούλια θα έπρεπε να κοιτάξουν στις χώρες τους πόσο καλή δουλειά κάνουν, πώς εμπλέκονται στις διάφορες διαδικασίες και όσον αφορά τα εθνικά τους προγράμματα. Μπορώ να σας πω ότι στη Φιλανδία συνεργαζόμαστε με την κυβέρνησή μας διαρκώς Ούτε ένα έγγραφο δεν φεύγει από το Φιλανδικό Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή που να μην το έχει εξετάσει το Φιλανδικό μας Κοινοβούλιο και να μην το έχει συζητήσει. Οι περισσότεροι από εμάς λοιπόν μπορούν αυτή τη στιγμή να πάμε στις χώρες μας και να δημιουργήσουμε συστήματα που μελετάει και το Συμβούλιο με δημοκρατικό τρόπο. Όπως πιστεύω τα περισσότερα ή όλα τα εθνικά κοινοβούλια υποστηρίζουν τις κυβερνήσεις τους και αντιστρόφως. Αυτό αφορά και το ζωτικό ζήτημα του προπολογισμού. Το δεύτερο που ήθελα να πω, όσον αφορά την οικονομική πολιτική, δεν μπορεί να εξετασει μόνο τη δημοσιονομική βιωσιμότητα εις βάρος ε, των υπόλοιπων σημαντικών στόχων όπως της απασχόλησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής σταθερότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο πλαίσιο του εξαμήνου και των εθνικών προϋπολογισμών. Να σας υπενθυμίσω ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Είναι δεσμευτικό σε ολόκληρη την ε, Ένωση. Όλη η νομοθεσία θα πρέπει να συντάσσεται και να εφαρμόζεται έτσι ώστε να διασφαλίζει τα κοινωνικά δικαιώματα που διασφαλίζει η συνθήκη αυτή. Και τρίτον, πιστεύω ότι η νέα η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα όλα τα επίπεδα των εθνικών προπολογισμών είναι η ε, φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή. Ε, τα ζητήματα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου θα αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της φοροαποφυγής. Ευχαριστούμε μιλητής πριν απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Καλτέρα από την Ισπανία. Να ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αυτό που ζούμε είναι μια κρίση σοβαρή οικονομικής ανάπτυξης που ε, καταργεί θέσεις απασχόλησης, αυξάνει το έλλειμμα και το χρέος τελικά και όχι το αντίστροφο. Στην περίπτωση της Ισπανίας είναι προφανές. Όταν άρχισε η κρίση η Ισπανία είχε πλεόνασμα και πολύ χαμηλό δημόσιο χρέος. Λοιπόν, η κρίση μας οδήγησε εδώ. Και ε, τα αποτελέσματα είναι όλο και χειρότερα κύριε Επίτροπη και για την Ισπανία και την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 2012 η Ισπανία 1,3% έπεσε το ΑΕΠ και χάθηκε 5% ε, από τις απασχόλησεις και ο πολλαπλασιαστής όλο και αυξάνεται. Τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, όχι μόνο για την Ισπανία και για την υπόλοιπη Ευρώπη. Τι μας ανησυχεί εμάς. Βλάπτονται οι δυνατότητες ε, της ανάπτυξης της οικονομίας για το μέλλον και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η Ισπανία έχει λάβει μέτρα πάρα πολύ βαθιά. Εγώ ανήκω στην αντιπολίτευση, ανεξάρτητα από το αν συμφωνώ ή όχι, κάνουμε μια υποτίμηση ανταγωνιστική. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετρία από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα για να υπάρξει μεν η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά μην οδηγεί σε χειρότερα δράματα. Αυτό πώς λύνεται. Εμπειρικά έχουμε αποδείξει πως η λιτότητα όλο και περισσότερο προκαλεί πιο αρνητικά προβλήματα και αποτελέσματα. Ένα είναι ο δρόμος. Επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις, το είπαν εδώ πολλοί συνάδελφοι. Επένδυση, μόνο έτσι θα βγούμε από την κρίση, αύξηση των επενδύσεων. Ούτε οι οικογένειες μπορούν να το κάνουν, ούτε επιχειρήσεις ε, με τη διαδικασία αυτή που ε, υπάρχει της λιτότητας. Αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο και σε εθνικό θα πρέπει να τονωθούν, να ευνοηθούν οι ε, επενδύσεις σε παραγωγική βάση για να επανέλθει στο δρόμο της ανάπτυξης η Ευρώπη. Νομίζουμε ότι υπάρχει χώρος γι' αυτό. Όλο και περισσότεροι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Ένα τελευταίο παράδειγμα. Η Κριστίν Λαγκάρτ, επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, πρόσφατα δήλωσε ότι είναι σχεδόν αδύνατο εμείς να επιστρέψουμε να αποπληρώσουμε τα χρέη μας αν δεν υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας. Και πρόσθεσε η κυρία Λαγκάρτ ότι θα πρέπει να γίνεται χωρίς αποκλεισμούς. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερος χρόνος για την ε, δημοσιονομική εξυγίανση και δυνατότητα παραγωγικών επενδύσεων για να επανέλθει η ανάκαμψη και η ανάπτυξη της οικονομίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και για την κατανόησή σας ότι τώρα ε, κάπως θα πρέπει να συμπιέσουμε το χρόνο και θα απαντήσει στις ερωτήσεις τώρα ο Επίτροπος κ. Ρέν. Thank you. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για την ε, πολύ ουσιαστική και σοβαρή συζήτηση που αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θα ήθελα να απαντήσω ομαδικά στις απαντήσεις, στις ερωτήσεις, ε, διότι είναι ο μόνος τρόπος να προλάβουμε. Άλλωστε το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να, να εξετάσουμε τα θέματα αναλυτικά. Θα ήθελα καταρχήν να ε, απαντήσω στον Λόρδο Χάρισον από τη Βουλή των Λόρδων. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ επικοδομητική Βρετανική συμβολή στην Ευρωπαϊκή Συζήτηση. Μου θυμίζετε ένα γεγονός ε, που έχει συμβεί εδώ και κάποια χρόνια. εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 1995 ήμουν Ευρωβουλευτής στην ε, Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και είχαμε μια συνάντηση με την αντίστοιχη Επιτροπή της Βουλής των Λόρδων. Στόχος ήταν να συζητήσουμε τα θέματα που σχετίζονταν με την τότε επικείμενη διακυβερνητική διάσκεψη στο Άμστερνταμ 1996-1997. Εμείς λοιπόν συναντηθήκαμε με τη Βουλή των Λόρδων. Ε, κάποια στιγμή δύο Λόρδοι άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους ηλικία 80 και 85 ετών αντίστοιχα. Και ο ένας έλεγε στον άλλον ότι εσύ φταίς που δεν συμμετέχουμε στην ε, διακυβερνητική διάσκεψη. Εσείς ε, λοιπόν αναφέρεστε στο 96, στο 1957, όχι. Μιλούσαν για την ε, διακυβερνητική διάσκεψη του 1951 και κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον γιατί δεν συμμετείχε τότε το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρώπη. Μπορεί οι λόγοι που δεν συμμετείχε το Ηνωμένο Βασίλειο τότε να έχουν ακόμα κάποιο, κάποιο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω τι ανησυχίε σα σχετικά με την ενιαία αγορά, σχετικά με τη μείωση τη γραφειοκρατία, ε, σχετικά με την πρόθεση του ελεύθερου εμπορίου. Ταυτόχρονα όμω, θα ήθελα να πω στον Πρωθυπουργό Κάμερον ότι δεν χρειάζεται κανείς να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αλλάξει το πολιτικό θεματολόγιο. Μπορεί κανείς να συνεργαστεί ε, με τα άλλα κράτη-μέλη εντός της Ευρώπης ως μέρος της κοινότητας στην οποία συμμετέχει κανείς. Αν ήμουν εγώ Βρετανός, θα προτιμούσα το Ηνωμένο Βασίλειο να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι και να ε, συμμετέχει στις αποφάσεις ε, παρά ε, να κάθεται στο πάγκο. Κανείς δεν έβαλε ποτέ γκολ από το πάγκο. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με το αίσθημα ιδιοκτησίας και την εθνική κυριαρχία που αναφέρθηκαν από πολλούς ε, συμπεριλαμβανομένου του κυρίου Φρέντο, του Μαρίνη, την κυρία Γκούλτα, τον κύριο Σέρβες και άλλους. Σας ακούω, ακούω αυτά που λέτε, τα καταλαβαίνω και συμφωνώ πολύ με τη σημασία του να υπογραμμίσουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε το αίσθημα ιδιοκτησίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου από τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια. Δύο πράγματα θα ήθελα να πω εδώ. Το ΣΥΚΣΠΑΚ, η οι των έξι νομοθετικών μέτρων που έχουν ενισχύσει την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη ε, ήταν νομοθέτημα όλων σας και τα 27 κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν ε, ε, τη δέσμη αυτή μετά από προσεκτική εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρασαν μήνες διαπραγματεύσεων και προσεκτική εξέταση των θεμάτων. Ο ρόλος της Επιτροπής τώρα λοιπόν είναι να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους κανόνες αυτούς, τους οποίους εγκρίνατε εσείς. Και περιμένουμε κάθε κράτος μέλος και κάθε κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σεβαστεί τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις και να κάνει αυτά που διδάσκει, δηλαδή να ε, σεβαστείτε την οικονομική διακυβέρνηση και τους κανόνες που ε, υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο του ΣΥΚΣΠΑΚ. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν τη βιωσιμότητα της, ε, των δημοσιονομικών απαιτείται αυτό. Το άλλο θέμα είναι ότι εμείς εξετάζουμε το θέμα αυτό από πλευρά τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εταιρική σχέση με τα κράτη-μέλη, με τα κοινοβούλια τους και οι πολιτικέ συστάσεις μας στόχο έχουν να βοηθήσουν κάθε κράτος μέλος να ξεπεράσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ε, να εξαλείψουμε τα σημεία συμφόρησης ε, και να επιτρέψουμε τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν με αντικειμενική ανάλυση της κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη και φροντίζουμε να παρέχουμε τις καλύτερες πολιτικές σύμβουλες με στόχο την αύξηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης. Κατόπιν είχαμε μια τρίτη ομάδα ερωτήσεων από διάφορους βουλευτές που είχαν να κάνουν ε, με ε, την δημοσιονομική εξυγίανση και το θέμα των δημοσιονομικών πολλαπλασιαστών, ε, τις ε, επιπτώσεις ε, δηλαδή διαφόρων μέτρων στην οικονομική ανάπτυξη. Και κάποιοι είπαν ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στα συμπτώματα αλλά και στις αιτίες της κρίσης. Ε, συμφωνώ απολύτως. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις αιτίες της κρίσης που είναι η οικονομική ανισορροπία τις μεγάλες ε, και ε, μη βιώσιμες οικονομικές ανισορροπίες ε, που προέκυψαν από το 2000 μέχρι περίπου το 2008. Αυτή είναι η πραγματική αιτία και γι' αυτό θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και γι' αυτό πρέπει να επιφέρουμε ισορροπία στην ευρωπαϊκή οικονομία και θα πρέπει και οι χώρες της Νότιας Ευρώπης ε, και οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης ε, να συμβάλλουν ώστε να έχουμε μια πιο γρήγορη επιστροφή στην ανάκαμψη και την αύξηση της απασχόλησης. Πρέπει να πω όμως ότι μερικές φορές ένα σύμπτωμα γίνεται αιτία. Και ενώ εδώ ότι ενώ λέμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της κρίσης, αυτό είναι απόλυτα σωστό, Ταυτόχρονα όμως δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας στα συμπτώματα της οικονομικής κρίσης, την ανεργία ή την απαιτούμενη δημοσιονομική εξυγίαση, τη μη βιωσιμότητα ε, των, ε, ε, των δημοσιονομικών. Και μελέτησα πολύ προσεκτικά την έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που αναφέρθηκε ε, είναι του Ολιβιέ Μπρανσάρτ, ε, του οποίου τα βιβλία διάβαζα όταν ήμουν φοιτητή. Ε, είναι και του νέου ερευνητή Ντάνιελ Λί. Είναι μια εξαιρετική έρευνα, εξαιρετικής ποιότητας. Στο έργο αυτό η Μπλάνσαρτ και Λί προειδοποιούν κατά της ερμηνείας των συμπερασμάτων τους ε, σχετικά με την εξεύρυνση τρόπου επίλυσης της ε, κρίσης. Γιατί, ε, διότι η Δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστέ ενδιαφέρουν από χώρα σε χώρα και εξαρτώνται από το γενικό οικονομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει λοιπόν ένα κανόνα που να μπορεί να εφαρμοστεί στο κάθε πλαίσιο και γι' αυτό η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ε, διαφοροποιημένης ε, δηλαδή εξυγίανσης ε, είναι η πιο κατάλληλη. Και θα πρέπει να πω εδώ ότι τα εμπειρικά στοιχεία που έχουμε μας δείχνουν ότι παρότι η εξυγένση σε κάποιες περιπτώσεις ε, οδήγησε σε κάποια προβλήματα δεν ε, σημαίνει ότι η διαφορετική λύση θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Ειδικά σε χώρες ε, με μεγάλο δημοσιονομικό χρέος Ε, θα είχαμε μεγάλα προβλήματα που θα αντιστάθμιζαν ε, την, ε, τα αποτελέσματα μιας πιο ήπιας μεταρρύθμισης. Ακόμα στις περιπτώσεις όπου οι αγορές δεν θα είχαν τη διάθεση να χρηματοδοτήσουν την, το, το δημοσιονομικό κρέας. Σκεφτείτε παρακαλώ την Ιταλία το φθινόπωρο του 2011 ανάμεσα στον Αύγουστο και τον Νοέμβριο του 2011. Η Ιταλία είχε δεσμευτεί στα τέλη του καλοκαιριού ε, να εξηγιάνει τα δημοσιονομικά της ε, και για να διευκολύνει ε, την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις δευτερεύουσες αγορές. Αυτό έγινε, παρενέβη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κατάσταση για λίγο άρχισε να βελτιώνεται. Τι έγινε μετά η κυβέρνηση Μπερλουσκόνη αποφάσισε να μην σεβαστεί τις δεσμεύσεις της. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Στέρεψαν ε, οι πόροι και ε, ε, σταμάτησε η ανάπτυξη και τελικά οδηγήθηκε σε πολιτικό αδιέξοδο η Ιταλία. Ο Μάριο Μόντι κατόπιν κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση. Και τέλος, ε, καθότι μου δείχνουν κίτρινη κάρτα, έχει τελειώσει ο χρόνος. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι η σημερινή συζήτηση ήταν πολύ χρήσιμη υπό την έννοια ότι δεν είδαμε το χάσμα βορρά και νότου που δυστυχώ βλέπουμε πολύ συχνά ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Με απασχολεί πολύ το πολιτικό χίσμα που υπάρχει ε, ανάμεσα στην ε, λεγόμενη κουλτούρα της σταθερότητας που υπάρχει στο Βορρά και στο Νότο, διότι ε, αυτά είναι ε, απλοϊκές ε, παρουσιάσεις της κατάστασης, καρικατούρες. Δεν υπάρχει μια χρυσή λύση στην κρίση αυτή. Δεν μπορούμε να τη λύσουμε μόνο με την δημοσιονομική πειθαρχία, διότι αυτό θα πνίξει την ανάπτυξη ούτε μπορούμε να τη λύσουμε μοιράζοντας ε, τους κινδύνους, διότι έτσι θα οδηγηθούμε σε υψηλό ηθικό κίνδυνο. Ε, γι' αυτό θέλουμε να γεφυρώσουμε τις δύο αυτές κουλτούρες και να ανοικοτομήσουμε την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, να έχουμε μια ένωση σταθερότητας με αυξημένη ευθύνη και αυξημένη αλληλεγγύη εγώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια τέτοια ένωση θέλουμε να οικοδομήσουμε και βασιζόμαστε στη δική σας υποστήριξη, διότι αυτή είναι η πραγματική βάση για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, αυτά που ζητάνε δηλαδή οι πολίτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια ωραία παροιμία που λέει δεν επιβραβεύεται η αρχαία, αλλά ε, μόνο ε, η διάρκεια και η αντοχή. Και αυτό θέλουμε να αντέξουμε. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας και για την υπομονή σας ε, και θα ήθελα να παραδώσω τώρα την Προεδρία στον κύριο Λαμασούτ, Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, για να μπούμε στην ειδική συζήτηση τώρα για τον προϋπολογισμό. Ευχαριστώ.